After Gesine start, I think. Ναι, και είναι εδώ η κυρία Μάσιναρ, μπορούμε να ξεκινήσουμε. Ξέρω ότι είχατε μια συνεδρία σκιωδών. Πολύ σημαντική. Για τα ποδήλατα, έτσι, το δεχθήκατε. Μπράβο και ευχαριστώ πολύ. Δεύτερο δώρο γενεθλίων από εσά για μένα. Λοιπόν, ξεκινάμε και έχουμε καταρχάς τις αποφάσεις της συνεδρίας των συντονιστών, σας τις διανύμαμε. Εάν μέχρι σήμερα το απόγευμα στις 6.30 δεν έχετε αντιρρήσεις, εγκρίνονται αυτές οι επιλογές των συντονιστών και από την Επιτροπή. Προχωρώ τώρα στην παρουσίαση της μελέτης για τις συνέπειες της ε, χρήσης των βιοκαυσίμων στις μεταφορές και το περιβάλλον. Ο κύριος Δεσάντη, η κυρία Μαρέλη είναι εδώ για μια παρουσίαση από το Κοινό Κέντρο Έρευνας Ινστιτούτο Ενέργειας Μεταφορών της ΙΣΠΡΑ. Θα μας παρουσιάσουν μια έκθεση την οποία έχει ζητήσει από το Πόλη Department η Επιτροπή μας ήδη πριν από τρία χρόνια, ογκοβέστατη όπως βλέπετε. Και δίνω το λόγο τώρα για την παρουσίαση στους προσκεκλημένους μας. Ποιος θέλει να ξεκινήσει. Ευχαριστώ πολύ κύριε Κράμερ. Καλησπέρα σε όλους. Πριν επισέλθουμε στις επιστημονικές λεπτομέρειες, επιτρέψατε μου να σας πω κάποια προσαγωγικά για αυτή τη μελέτη. Αυτή η μελέτη, όπως μπορείτε να διαπιστώσετε από τον τίτλο, αφορά τις επιπτώσεις των βιοκαυσίμων που ό,τι μπορεί να υπάρξει ή γίνεται να υπάρξει τέλος πάντων σε διάφορους τρόπους ε, μεταφοράς και τη σχέση με την ανάπτυξη της γεωργίας στην Ευρώπη. Οπότε θα, είπαμε ότι θα ε, μαζέψουμε όλα τα δεδομένα, τις αναλύσεις που έχουν γίνει και από όλες τις ε, πηγές ΩΣΑ και όλες. Για να δούμε επομένως τι επιπτώσεις υπάρχουν στου διάφορου κλάδου οικονομίας στα βιοκαύσιμα. Αυτό ήταν ο στόχο τη Είμαι επικεφαλή του Ιδρύματος ε, του, ε, του για τις επιστημονικές έρευνες, αλλά και η κυρία Λουίζα Παρέλη είναι η υπεύθυνη για συγκεκριμένη μελέτη. Προχωρούμε. Λέμε ότι αυτή η Γενική Διεύθυνση, η GRC, είναι η αρμόδια για να ε, διεξαγάγει την έρευνα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αυτή την έρευνα, και επομένως έτσι έχουμε τεκμηρίωση επιστημονική για τη χάραξη των πολιτών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Βλέπετε, επομένως, τι κάνουμε. Ε, έχουμε εστιάσει την δραστηριότητά μας σε κάποια βασικά θέματα όσον αφορά το θεματολόγιο του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όποτε χρειάζεται. Ενέργεια και μεταφορές τώρα. Όπως βλέπετε το Ίδρυμά μας έχει πάρα πολύ ευρία γκάμα δραστηριοτήτων και τώρα μιλούμε για τα βιοκαύσιμα. Εν προκειμένου και στο παρελθόν, βέβαια έχουμε κάνει διάφορες μελέτες και κατά αυτόν τον τρόπο προσπαθούμε να εντοπίσουμε το πώς γίνεται η χρήση της ενέργειας σε σχέση με το φαινόμενο του θερμοκηπίου πάλι συνδέοντά το με τα διάφορα είδη καυσίμων. Προσπαθούμε να έχουμε μια μεθοδολογία ξεκάθαρη και διάφανη. Να λάβουμε επομένω υπόψη τη χρήση τη ενέργεια και τη θερμοκηπίου σε όλο τον κύκλο ζωή του, του καυσίμου. Από την άντλησή του λοιπόν, από την γεώτρηση βροσιπίν μέχρι το τέλο τη διαδρομή του. Και συνεργαζόμαστε βεβαίω και με την αυτοκινητοβιομηχανία αλλά και με τι πετρελαϊκέ εταιρείε. Ε, επίσης υπάρχει πρώτερα εμπειρία όσον αφορά τα βιοκαύσιμα. Οπότε για την οδηγία για την ποιότητα των καυσίμων, για την οδηγία για τη βιομάζα, για όλα αυτά τα νομοθετήματα ε, παρέχουμε την τεκμηρίωση. οπότε βλέπετε πως ε, αναλύσαμε τις τιμές τις σχετικές με, το, ε, με τα βιοκαύσιμα και τη βιομάζα. Και νομίζω ότι έχουμε συμβάλει αρκετά γιατί έχουμε δώσει για το ILOC ε, στοιχεία αντικειμενικά. Είναι δύσκολα, λεπτά θέματα, αλλά η εμπειρογνωμοσύνη μας νομίζουμε ότι έχει βοηθήσει στην ζήμωση στο πλαίσιο του ILOC για την βιοενέργεια, για τα δάση κλπ. Και όπως διαπιστώνετε, το Ίδρυμά μας έχει αναπτύξει προγνωμοσύνη και γνώση για όλα αυτά τα σημαντικά ζητήματα, τα μας στη συγκεκριμένη περίπτωση και τη χρήση τους. Ολοκληρώνοντας θέλω να πω ότι αυτή η μελέτη τι αφορά. Πρώτα πρώτα. Υπάρχει μια σύμβαση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το Δεκέμβριο του 12. Και τα αποτελέσματα είναι το έγγραφο και η ανάλυση το Δεκέμβριο του 13. Ένα χρόνο μετά. Προσθέσαμε τα αποτελέσματα τον Απρίλιο του 2014. Ήδη επομένω σε αυτή την ίδια αίθουσα έχει γίνει η παρουσίαση τη μελέτη πριν από ένα χρόνο. Και έχουν την τελική εκδοχή του κειμένου και όλε τι παρατηρήσει του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και από τι διάφορε γενικέ ε, διευθύνσει τον Ιούλιο του 2014. Οπότε από τότε ε, είναι δημοσία και διατίθεται για όποιον θέλει η τελική μορφή της έκθεσης. Πάμε τώρα στο επιστημονικό τμήμα της παρουσίασης. Σας υπενθυμίζω πάντως τους στόχους της μελέτης. Όπως είπαμε θέλουμε να αναλύσουμε τις επιπτώσεις. Δηλαδή, τι γίνεται με την ασφάλεια της προμήθειας. Πώς δηλαδή τα βιοκάψιμα μπορούν να δώσουν περισσότερες επιλογές για τις ε, πηγές όσον αφορά την ασφάλεια της προμήθειας. Ποια είναι τα αποτελέσματα όσον αφορά την απασχόληση. Δημιουργεί νέες θέσεις ε, εργασίας. Υπάρχουν θετικές ενεργές εκτόσεις για την οικονομία. Πολύ σημαντικό σημαίνει συγκυρία. Ε, επίσης, τις ε, επιπτώσεις όσον αφορά τη γεωργία και τις αγροτικές τιμές και τι γίνεται με την ε, χρήση της γης. Πώς δηλαδή η πολιτική επηρεάζει την χρήση των γεωργικών γεών αλλά και των μη γεωργικών και την μεταβολή στην χρήση επίσης αυτών των γεών. Επίσης, τι γίνεται όσον αφορά την καταπολέμηση των εκπομπών που δημιουργούν το φαινόμενο του θερμοκηπίου. Επίσης, τι γίνεται όσον αφορά την τεχνολογία, δηλαδή το πώς τα διάφορα βιοκάψιμα συμπεριφέρονται. Δεν είναι όλο το ίδιο και πώς η τεχνολογία θα εξελιχθεί στο μέλλον. Γιατί πάμε από την πρώτη γενιά στην δεύτερη. Να δούμε ποια είναι τα πλεονεκτήματα, ποια είναι η φραγμή από την τεχνολογία επιστημονικής αλλά και οικονομικής φύσεως. Και να δούμε τι πολιτική χρειάζεται ώστε να μπορέσουμε να έχουμε κάποιο είδους σταθερό, γερό, επενδυτικό πρόγραμμα. Όσον αφορά τη δεύτερη ή τρίτη γενιά βιοκαυσίμων. Όπως βλέπετε έχουμε αναλύσει πάρα προνοιδών επιπτώσεις. Άρα τώρα για να δούμε η κυρία Μορέλη τι έχει να μας πει για τα καθέκα στον σημείο της μελέτης. Ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα σας. Θα προσπαθήσω να κάνω κάποιες σύντομες παρεμβάσεις για τα βασικά ευρήματα της μελέτης και θα αφήσω και χρόνο για να τα συζητήσουμε μετά. Ακολουθώντας τα όσα μόλις εξήγησε ο κύριος Ντεσάντη, έχουν να κάνουν με την ασφάλεια των εφοδιασμού που αποτελεί έναν από τους πυλώνες πολιτικές μας από το 2009. Όντως ε, βοηθούν στην διαφοροποίηση των πηγών για τα καύσιμα μεταφορών και σύμφωνα με τους υπολογισμούς που κάναμε και από την USDA αλλά και από την CONCAO που είναι ο σχετικός, η σχετική ένωση των Ευρωπαίων ε, κατασκευαστών το 5,1 το 2011 των καυσίμων ήταν βιοκαύσιμα. Θα πρέπει να δούμε τι είδε η Eurostat. Το 2013 είπε ότι μόνο το 4,8% των καυσίμων είχαν υποκατασταθεί από βιοκαύσιμα στην Ευρώπη. Τώρα για το 2020 τι λένε οι προβλέψεις, 10 δις λίτρα βενζίνης θα εξοικονομηθούν και σύμφωνα με τη νέα πολιτική που προτείνουμε μπορεί αυτό να αλλάξει μια και υπάρχουν αυτές οι οροφές στην ε, παραγωγή βιοεθανόλης ε, και βιοδίζελ πρώτης γενεάς. Τώρα, αρνητικό αρνητικός ή θετικός αντίκτυπος στην τοπική οικονομία. Γενικά είναι μάλλον θετικός αντίκτυπος και κυρίως στις περιοχές της αγροτικής της υπαίθρου. Αυτό θα πρέπει να εξορροπηθεί με την αρνητική επίπτωση που είναι η αυξημένη φορολογία λόγω του υψηλότερου κόστου παραγωγής των βιοκαυσίμων. Οι προβλέψεις για άμεσες θέσει εργασίας στον κλάδο είναι το 2011 120.000 νέες θέσει εργασίας όμως, αυτό ισχύει αν δεν λάβει υπόψη την επιπλέον φορολόγηση και το επιπλέον κόστος. Στις μελέτες που το κάνουν ε, αυτό βλέπουμε πως τα πλεονεκτήματα αυτά έχουν επιτευχθεί με κάποιες απώλειες σε άλλους κλάδες, οπότε τελικά υπάρχει ένα μικρό θετικό πρόσημο, καμιά φορά και αρνητικό στον υπολογισμό. Κόστος. Η στήριξη των βιοκαυσίμων στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι από το 7 μέχρι 8 ε, δις ευρώ το 2011, δηλαδή 14 με 17 ευρώ ανά Ευρωπαίο. Για ποιο λόγο υπάρχει αυτό το κόστος, γιατί τα βιοκαύσιμα στην παραγωγή τους είναι πιο ακριβά. Πιο ακριβά από το παραδοσιακό δίζελ και βενζίνη, αλλά τα βιοκαύσιμα πολλούνται ε, στην ίδια τιμή στα βενζινάδικα, στην Αντλία δηλαδή, οπότε υπάρχουν φόροι κατανάλωσης, φόροι ειδικοί και άλλοι φόροι που δημιουργούν αυτό το επιπλέον κόστος. Τελικά, σε 17% υψηλότερο κόστος παραγωγής από ό,τι τα παραδοσιακά καύσιμα. Η γεωργία. Τα βιοκαύσιμα επηρέασαν σε μεγάλο βαθμό ε, τις ανάγκες ε, για ε, φυτικά έλαια στην Ευρώπη. Και αυτή η αυξημένη απέτηση αντιμετωπίστηκε με εισαγωγές από την Ινδονησία και, του, και το μπαλί φινικελαίου και από τη Βραζιλία και αυτό γιατί έχουν τη δυνατότητα να κάνουν αυτή την καλλιέργεια σε ε, εδάφη ε, παρθένου δάσους στις χώρες τους και αυτό όμως οδήγησε σε αυξημένα σε εκπομπές λόγω αυτής της καλλιέργειας ε, να σας πω πως το ένα λίτρο φινικέλου που χρησιμοποιείται για το βιοντίζελ ε, αφαιρείται από το λάδι, το φινικό ε, δηλαδή που είναι διαθέσιμο ως τρόφιμο. Αυτό όμως χρησιμοποιείται για να υποκαταστήσει το κρανβέλο που χρησιμοποιούμε για τα βιοκαύσιμα στην Ευρώπη. Τα βιοκαύσιμα λοιπόν σημαίνουν πως υπάρχει αυξημένη ζήτηση κάποιων καλλιεργειών Βλέπετε με τη μαύρη γραμμή τιμή πετρελαίου, αργού πετρελαίου, πράσινο, ε, μπλε και ε, κόκκινο είναι τα τρία φυτικά έλαια ε, και βλέπετε ότι δεν υπήρχε καμία σχέση μεταξύ της πορείας αυτών και του αργού και μάλιστα πως υπήρχε μια μείωση τιμή μέχρι το 5, από το 2005 και μετά η στιγμή που μπήκαν αυτά τα έλαια στην αγορά, αυτά τα τέσσερα αγαθά έχουν παρόμοιες πορείες τιμών. Ε, βλέπουμε λοιπόν πως υπάρχουν συνέπειες από την είσοδο των βιοκαυσίμων στην αγορά ε, καυσίμων ε, γενικότερα. Για την εθανόλη είναι πιο δύσκολο να κάνουμε παρόμοια αξιολόγηση γιατί η αγορά σακάριων και δημητριακών είναι πολύ μεγαλύτερη από αυτή για τα φυτικά έλαια και η νέα παραγωγή εθανόλης είναι πολύ μικρότερη σε όγκο από αυτή του βιοντίζελ. Άρα λοιπόν στην παγκόσμια αγορά δημητριακών είναι δυσκολότερο να εντοπίσουμε πώς επηρεάζει η ζήτηση εθανόλης στις τιμές. Πάντως, είχαμε το ίδιο φαινόμενο πως είχαμε στις τιμές για το βιοντίζελ και τα φυτικά έλαια. Δηλαδή, καλα, για το καλαμπόκι, τον αρβόστο δηλαδή, εδώ έχουν παρόμοια πορεία με την πορεία του αργού και από το 2005 και μετά αυξάνεται η τιμή τους από τη στιγμή δηλαδή που μπαίνουν αυτά στην αγορά. Για τη χρήση γης και τις συνέπειες εκεί, 5,7 δύο γης χρησιμοποιήθηκαν παγκοσμίως για να, για να καλλιεργηθούν αυτά τα βιοκαύσιμα που χρησιμοποιούμε στην Ευρώπη. Το 2010 το μερίδιο των βιοκαυσίμων ήταν το 4,27% για τις μεταφορές. Η πλειονότητα αυτής της χρήσης γης στην Ευρώπη και το 43% προέρχεται από το εξωτερικό. Αυτό το 5,7 εκτάρια αντιστοιχεί σε 5 περίπου 100% της αρρώσιμης γης. Αυτή η αυξημένη απέτηση για καλλιεργείς μπορεί να προκαλέσει μια μετακίνηση ε, παραγωγής ε, τέτοιων καλλιεργιών για τρόφιμα προς άλλες περιοχές. Άρα έχουμε λοιπόν μια έμεση αλλαγή χρήσης γης το iLook και αυτές οι εκπομπές δεν λαμβάνουν υπόψη στην νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ακόμα. Γίνεται βέβαια μεγάλη πολιτιστική συζήτηση, αλλά τα συμπεράσματα όλων των επιστημόνων είναι πως τελικά το μέγεθος των εκπομπών αυτών ε, είναι αβέβαιο, πάντως η επιστήμη αποδεικνύει πως τελικά στις εκπομπές, στην εξοικονόμηση εκπομπών ε, αερίου του θερμοκηπίου αυτές οι εκπομπές ILUC έχουν μεγάλη επίπτωση. Για να τις αξιολογήσουμε χρειαζόμαστε ένα οικονομετρικό μοντέλο για να λάβουμε υπόψη όλους τους συσχετισμούς μεταξύ αγορών με προβλέψεις για το μέλλον. Για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να σας πω μόνο πως θεωρήσαμε ως μοντέλο αναφοράς τη μελέτη του Διεθνούς η ε, Ινστιτούτο Ερεύνης για τα ε, τρόφιμα και εδώ στον πίνακα λένε πως οι εκπομπές αερίου θερμοκηπίου που δημιουργούνται από τα iLook, κυρίως για τα δημητριακά ζάχαρα και τα φυτικά έλαια, είναι τα εξής. Βλέπετε λοιπόν πως δημοκρατικά ζάχαρη για την εθανόλη έχουν πολύ χαμηλότερη επίπτωση από αυτές του βιοντίζελ και ένα μεγάλο τμήμα αυτών των υψηλότερων εκπομπών εξηγείται από το γεγονός πως ε, έχουμε την καλλιέργεια φινικελαίου σε ε, τις σε πολύ συγκεκριμένε και μικρές περιοχές του κόσμου. Από εκεί προκύπτουν. Και μπορούμε να το λάβουμε υπόψη όταν χρειαστεί να έχουμε καλύτερες επιδόσεις και αποδόσεις με την καλλιέργεια βιοντίζελ. Έχουμε διάφορα οικονομικά μοντέλα και πρόσφατα λάβαμε και δύο μελέτες που έδωσαν προσωρινά στοιχεία, τα οποία συμπεριλαμβάνουμε και εμείς στην έκθεση, όπου βασιζόμαστε σε ιστορικά στοιχεία και επιβεβαιώνουμε αυτές τις τάσεις, τις εκπομπές iLook που προέκυψαν και από τα οικονομητρικά μοντέλα. Για τις ε, εξοικονόμηση εκπομπών αερίου θερμοκηπίου, να σας πω πως μόνο ε, θα προκύψουν εάν δεν λάβουμε υπόψη κομπές άιλουκ. Αν όμως τις συμπεριλάβουμε, για παράδειγμα έτσι όπως υπολογίστηκαν προηγουμένως, τότε δεν εξοικονομούμε καθόλου για το βιοντίζελ και πολύ μικρότερες εξοικονομήσεις στο θέμα της εθανόλης. Εκεί υπάρχει δυναμικό αυξημένης ε, εξοικονόμησης χρησιμοποιώντας και στην εξίσωση τα Outlook, θα μιλήσω γι' αυτό αργότερα. Σας έδειξα λοιπόν τι γίνεται με τις εκπομπές από τα περισσότερα βιοκαύσιμα, με γαλάζιο έχω τις άμεσες εκπομπές και με σκούρο μπλε τις έμεσες. Βλέπετε λοιπόν πως για το βιοντίζελ δεν έχουμε εξοικονόμηση, αλλά στην πραγματικότητα αύξηση εκπομπών, εάν συγκρίνουμε με το τι γίνεται όταν χρησιμοποιούν ορυκτά καύσιμα έχουμε δυνατότητα για περαιτέρω Για παράδειγμα, υποπροϊόντα ε, τα οποία ε, ε, συμπαράγονται εάν κάνουμε συμπαραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας ή θερμότητας. Επίσης μπορούμε να απαγορεύσουμε σε τριφοειδή εδάφη να έχουμε καλλιέργεια φινικελαίου Επίσης, μπορούμε να αποφύγουμε αυτές τις εκπομπές ή να τις μειώσουμε αν τα βιοκαύσιμα ε, έρχονται από εγκαταλελειμμένη ή σε κακή κατάσταση γη, ε, με τον τρόπο αυτό μπορεί κανείς να αποφύγει τα προβλήματα ή να έχει, κάποιες ε, παράλληλες, να έχει κάποια παράλληλα πλεονεκτήματα, όπως για παράδειγμα χρήση υπολοιμάτων τροφίμων. Θα σας δείξω εδώ ένα πίνακα με το κόστος, παρόμοιο με αυτό που είδατε προηγουμένως. Βλέπετε λοιπόν πως η εξοικονόμηση διοξιδίου του άνθρακα με τα βιοκαύσιμα είναι δαπανηρό. Πάνω από 100 ευρώ ανά τόνο ε, διοξιδίου, πιο πολύ αν συμπεριλάβουμε και τα άλλο και το βιοδίζελ που είναι τα σκούρα μπλε τόξα. Δεν έχουμε καθόλου εξοικονόμηση έτσι κι αλλιώς, άρα είναι σχεδόν άπειρο το κόστος. Ε, επαναλαμβάνω, αν συνυπολογίσετε τα Προς το τέλος της παρουσίασης θα ήθελα να σας κάνω κάποιες προτάσεις για το προς τα πού μπορούν να κινηθούν τα βιοκαύσιμα. Στην πολιτική συζήτηση έχουμε μετακινηθεί περίπτωση προς τα βιοκαύσιμα δεύτερης ή τρίτης γενεάς, γιατί δυνάμει περιβαλλοντικά είναι πιο θετικά και έχουν και κάποια άλλα πλεονεκτήματα. Είναι αλήθεια πως εκεί έχουμε μεγαλύτερη εξοικονόμηση ε, εκπομπών ε, αερίων του θερμοκηπίου. Δηλαδή η παραγωγή των καυσίμων βασιζόμενη στη μεθοδολογία που ορίσαμε στην νομοθεσία είναι μειωμένη. Βλέπετε εδώ τις τιμές για, τα, για την θερμότητα, για την ηλεκτρική ενέργεια, όπως επίσης και τα καύσιμα μεταφοράς. Κάνουμε τις συγκρίσεις και οι εκπομπές είναι πάντα και σε κάθε περίπτωση χαμηλότερες από αυτές των ορυκτών καυσίμων. Όμως, θα πρέπει να σταθούμε συνετοί τη στιγμή της αξιολόγησης, γιατί υπάρχουν και άλλες επιπτώσεις από τα δεύτερη γενιάς βιοκαύσιμα. Να κάνουμε ό,τι κάναμε και με τα έμεσα iLook, και να λάβουμε υπόψη ποιες είναι οι πιθανές έμεσες συνέπειες ε, στο περιβάλλον, στην οικονομία, στην κοινωνία. Χρήση υπολοιμάτων, για παράδειγμα, για την παραγωγή βιοκαύσιμα. Για να δούμε, είναι ανταγωνιστικά με άλλους κλάδους. Υπάρχουν ήδη χρήσεις αυτών των προϊόντων όπου απλώς ε, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα προϊόντα αυτά ως ε, καθαρά λιπαντική ε, ουσία. Πώς επηρεάζουν τον ευτροφισμό, τα ύδατα, τη ρήπανση του ατμοσφαιρικού αέρα και τι τύπος εξοικονόμησης αερίων γίνεται. Σας έδωσα κάποια παραδείγματα για κάποιες ζωοτροφές που προέρχονται από τη δασοκομεία, εκεί μειώνονται οι εκπομπέ αλλά μετά από πάρα πολλά χρόνια. Οπότε η θέση της ε, ε, ουδετερότητας εκπομπών δεν ισχύει. Επίσης, πώς επηρεάζεται η γη, τα εδάφη. Δεν λαμβάνεται αυτό υπόψη στη μεθοδολογία τη οδηγία. Τεχνικές, τεχνολογικές επιλογές. Για το βιομεθάνιο, για παράδειγμα μπορεί εκεί να έχει μεγάλες εξοικονομήσεις ε, στα, θερμο, στα αέρια θερμοκηπίου, αλλά με εσωτερικά χωνευτήρια. Αν όμως η κοπριά αφαιθεί σε ένα ε, ανοιχτό ε, χωνευτήριο, τότε εκτινάσονται οι εκπομπές. Αυτή τη στιγμή η πρόοδος που γίνεται στα βιοκαύσιμα δεύτερης γενιάς είναι πιο αργή από ό,τι περιμέναμε, γιατί οι τεχνολογίες λειτουργούν μεν, αλλά το κόστος εξακολουθεί να είναι εξαιρετικά υψηλό. Τι λέει η IEA. Το κόστος θα είναι συγκρίσιμο με αυτό των πρώτων γενεάς μόνο γύρω στο 2030. Έχουμε και πολλές ελπίδες για τα τρίτης γενεάς φύκια αλλά ακόμα είμαστε στη φάση της ε, εργαστηριακής μελέτης, οπότε ακόμα δυστυχώς τα φύκια δεν έχουν βγει στην αγορά. Οι φορείς λοιπόν θέλουν μια σταθερή πολιτική έτσι ώστε να μπορούν να επενδύσουν. Το συμπέρασμά μου είναι όπως βλέπετε και εσείς, πως είναι μόνο μία από τις εναλλακτικέ τα βιοκαύσιμα στο να μειώσουμε τις εκπομπές διοξιδίου στις ε, μεταφορές, αλλά είναι δαπανηρός τρόπος. Εκτός, ε, συγχωρείτε, εάν ιδιαίτερα να συγκριθούν με άλλες χρήσεις που μπορεί να έχει βιομάζα, για παράδειγμα, ηλεκτρική ενέργεια, θέρμανση κτλ. Θα πρέπει λοιπόν για τα προχωρημένα βιοκαύσιμα να δούμε ποια είναι τα πλεονεκτήματα και ποια είναι τα μειονεκτήματα που προσφέρουν πριν λάβουμε κάποιες αποφάσεις για το τι θα πρέπει να επιλέξουμε. Βιωσιμότητα, η οικονομική βιωσιμότητα της δεύτερης γενεάς θα επιτευχθεί πώς με μία εκτείναξη της χρήσης ή αν έχουμε κάποιες ε, οικονομικές λύσεις για τις ζωοτροφές ή αν υπάρχουν άλλα χημικά προϊόντα όπως έχουμε στα βιοδηληστήρια θα πρέπει η παραγωγή βιοκαυσίμων και τα βιοδηληστήρια να ε, χρησιμοποιηθούν μαζί με άλλες βιομηχανικές εγκαταστάσεις έτσι ώστε να έχουμε και άλλα βιοπροϊόντα, υλικά και καύσιμα για να έχουμε μεγαλύτερη ενεργειακή αποδοτικότητα και χρειαζόμαστε ένα πλαίσιο για να κινητοποιήσουμε τις επενδύσεις. Ο κλάδος λοιπόν ζητά έναν οικονομικό μηχανισμό πέραν αυτών που έχουν ήδη εφαρμοστεί ε, όπως το Horizon 2020 ή το NER 300, τα διαστροτικά ταμεία κτλ. Εκτός από τη μελέτη αυτή την οποία εμείς ε, ε, παραγγείλαμε, κάθε δύο χρόνια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναφέρεται στο Κοινοβούλιο για τις επιπτώσεις των βιοκαυσίμων όπως απαιτεί η οδηγία και πολύ πρόσφατα, πριν από μερικές μέρες, δημοσιεύσαμε την τελευταία μας αναφορά. Σας είπα πως Έχουμε σταθεί πολύ στο θέμα των προχωρημένων, εξελιγμένων ή δεύτερης γενεάς βιοκαύσιμα. Αυτό είναι κάτι που κάνουμε πολύ εμείς στο JRC. Και βλέπουμε και κάποιες άλλες εναλλακτικές λύσεις, έτσι ώστε να έχουμε ολόκληρη την εικόνα για τα νέα αυτά καύσιμα τα οποία βγαίνουν στην αγορά. Ευχαριστώ. Yeah, thank you very much for the presentation. Ευχαριστώ και εγώ την παρουσίαση. Παρακαλώ, ερωτήσεις. Μάλιστα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Δύο ερωτήσεις. Καταρχάς, ευχαριστώ θερμά για την έκθεση. Πολλοί θα τη μελετήσουν με μεγάλο ενδιαφέρον. Είναι πολύ αυτή στη Σουηδία, Φερρυπίνη, οι οποίοι θα ενδιαφερθούν ιδιαίτερως για τα χωρίσματά σας. Εγώ κατοικώ στην Βόρεια Σουηδία. Εκεί αποφασίσαμε να εξασφαλίσουμε μεταφορές χωρίς ε, ορυκτά καύσιμα μέσα στα επόμενα δύο χρόνια. Κοινότητες, περιφέρειες, δηλαδή επιδιώκουν τον ίδιο στόχο. Πώς μπορούμε όμως να τον εξασφαλίσουμε το στόχο αυτό. Έχουμε τις εξής διαπιστώσεις. Πρώτον, διαπιστώνουν οι κοινότητες, και κοινότητες, ότι μπορούμε να παραγάγουμε τα δικά μας βιοκαύσιμα. Έχουμε επαρκή ε, λίματα για να μπορέσουμε να τα μετατρέψουμε σε βιοκαύσιμα. Μπορούμε να κάνουμε τη λεγόμενη κομποστοποίηση από τα νοικοκυριά που έχει ξεκινήσει εδώ και αρκετά χρόνια, τουλάχιστον στη δική μου την ε, περιοχή. Και ναι, μπορεί να έχει σχετικά περιορισμένη έκταση, αλλά πάλι δίνει τη δυνατότητα σε τοπικό επίπεδο να γίνει αυτή η μετατροπή και επίσης δίνει και την αίσθηση ότι ε, ο, της ε, ιδιοποίησης του στόχου, ότι δηλαδή θέλουμε αυτή την, αυτό το στόχο να τον επιτύχουμε. Και βεβαίως θέλουμε να φτάσουμε στον χώρο των μεταφορών, αλλά τέτοιου είδους τοπικού χαρακτήρα δραστηριότητες αναπτύσσονται σε διάφορες περιοχές και έστω και χωρίς γενίκευσή τους μπορούν να δώσουν κάποια συγκεκριμένα αποτελέσματα. Στα δάση επίση, ξέρετε ότι η Σουηδία και η Φινλανδία κατέχουν τις μεγαλύτερες δασικές εκτάσεις της Ευρώπης και μπορούμε να πούμε ότι θα έχουμε και τα σχετικά, ε, τις σχετικές εκτάσεις παραγωγής βιοελαίων όταν γίνεται κοπή δέντρων αντικαθίστανται αυτά με αναδάσωση και έτσι γίνεται η ανανέωση των δασών. Άρα νομίζω ότι εδώ έχουμε μία δυνατότητα γιατί η βιομηχανία του χάρτου, παραδείγματι, διαπιστώνει πως μειώνεται η κατανάλωση χάρτου, άρα χρειάζεται να βρει λύσεις άλλες για να αξιοποιεί οικονομικά τα δάση. Εδώ μία λύση μπορεί να είναι η παραγωγή ενέργειας από τα δάση. Ε, μπορούμε να προβάλλουμε δηλαδή την ιδέα του βιοκαυσίμου από τις ε, δασικές εκτάσεις και νομίζω ότι πρέπει να επιδιώξουμε αυτό το στόχο από τα δάση να βλύσουμε μια επαρκή, έναν επαρκή ενεργειακό πόρο για όλη την Ευρώπη. Αυτό νομίζω πρέπει να το κοιτάξουμε. Εσείς τι γνώμη έχετε γι' αυτό. Ο πρόεδρος, ευχαριστώ. Βίρκουνεν. Μετά τη Σουηδία η, η Φιλανδία. Ευχαριστώ πολύ, πρόεδρε. Ευχαριστώ και τους επιστήμονες και ερευνητέ μας για την ε, παρουσίαση της έκθεσης. Ένα σχόλιο και δύο ερωτήσεις. Θα ήθελα καταρχάς σχολιάζοντας να σημειώσω αυτό που και ο κύριο Γιάννησεν και εγώ από τη Φινλανδία έχω, έχω να αναφέρω υψηλό επίπεδο χρήσης βιοκαυσίμων περί το 8% του βιοδίζελ του δίζελ θα πρέπει να προέρχεται από βιοκαύσιμα από φέτος. Το ποσοστό αυτό θα πρέπει να φτάσει στο 20% Πρέπει να αξιοποιηθούν οικιακά απόβλητα, υπόλοιπα τροφίμων κτλ. Για να έχουμε στο δυνατόν πιο μεγάλη αποτελεσματικότητα στη χρήση της ενέργειας. Εγώ θα ήθελα ως προς τα είδη των βιοκαυσίμων να σας ρωτήσω ποιο θα λέγατε ότι είναι το καλύτερο για το περιβάλλον, ποιο βιοκαύσιμο είναι πιο οικολογικό αλλά και οικονομικά πιο βιώσιμο. Επίσης, η ιδέα ανάπτυξης ε, βιοκαυσίμων δεύτερης και τρίτης γενιάς προχωράει με πολύ βραδείς ρυθμούς στην παραγωγή. τι είδους κενά υπάρχουν, τι αβεβαιότητες και πώς μπορούν να καλυφθούν. Οι στόχοι για τις κλιματικές αλλαγές του 2030. Φερρυπίνη δεν αναφέρουν τίποτα για τις μεταφορές και τα βιοκαύσιμα. Θα θέλαμε να βελτιώσουμε την αποτελεσματική ανάπτυξη αυτή τη δεύτερη και τρίτη γενιά. Τι έχετε να απαντήσετε, πώ μπορεί να εξασφαλιστεί αυτό. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Μάισνερ. Ευχαριστώ και εκ μέρου των φιλελευθέρων για τις παρουσιάσεις, ήταν πολύ συναρπαστικέ. Νομίζω ότι αν ήταν πιο φθηνό το βιοκαύσιμο θα το θέλανε όλοι. Εμεί τουλάχιστον στο Όφρο και κάνονται φήμησή μου εδώ έχουμε καταφέρει πάρα πολύ καλά αποτελέσματα. Βέβαια δεν μπορούν να τα καταφέρουν όλοι. Πρέπει να κοιτάξουμε και με προστασία του ε, περιβάλλοντος, της οικολογίας, να εξασφαλίσουμε βιοκαύσιμο με χαμηλές εκπομπές. Υπάρχουν διάφορες εναλλακτικές που μας ε, προτείνατε, κόστος, πρόσθετες εκπομπές, από τη χρήση της βιομάζας. Νομίζω ότι και εδώ θα συμφωνήσω με τον Σουηδό σοσιαλιστή συνάδελφο ότι μπορούμε να εξασφαλίσουμε και από τα δάση ε, υλικό, γιατί υπάρχει μια σειρά από απόβλητα των δασών, χωρίς να χρειάζεται να γίνει αποψήλωση ή κοπή δέντρων, που θα μπορούσε να αξιοποιηθεί για την παραγωγή βιομάζας. Ίσως όχι σε όλα τα κράτη της Ευρώπης όντως, αλλά τουλάχιστον στα σκανδιναβικά και βέβαια και η Γερμανία έχει αρκετά δάση, αρκετές δασικές εκτάσεις για το ήλοκ, για την έμεση δηλαδή χρήση γης. Έχουμε ξεκινήσει σε σχέση με την παραγωγή βιοκαυσίμων, βιοαερίου, ε, κάποιες προσπάθειες και αυτό σημαίνει ότι εκτάσεις αρρώσιμες έχουν φύγει από την παραγωγή τροφίμων για να αξιοποιηθούν για ε, βιοκαύσιμα. Αυτό όμως μπορεί να γίνει και συνδυασμένα, δηλαδή να γίνεται παραγωγή σιτηρών φερρυπίν, τα οποία και ως τρόφιμα αλλά και ως βιοκαύσιμα μπορούν να αξιοποιηθούν. Διπλή δηλαδή χρήση, διπλή χρήση. Και ερώτηση έχω την εξή. Για την τρίτη γενναία έχετε κάτι να πείτε. Τα φύκια τα έχετε λάβει υπόψη ω δυνατότητα, γιατί βέβαια τα φύκια τα βρίσκουμε μόνο στις θάλασσες, αλλά υπάρχει δυνατότητα. Και ξέρετε, ήμουνα σε μια δεξίωση της έρβας πριν από κάποιο διάστημα, που μιλούσε για τη δυνατότητα αξιοποίηση φυκιών για τις... Ε, ε, για τα βιο, ως βιοκαύσιμα. Το ίδιο ξέρω ότι έχει κάνει και η Boeing, εναλλακτική δηλαδή ε, μορφή καυσίμου για τις εναέρειες μεταφορές που προέρχεται από τα φύκια. Ε, μας λένε βέβαια ότι είναι ακόμα σε στάδιο ερευνητικό αυτό το σχέδιο. Υπάρχει δυνατότητα να δούμε και την οικονομική αξιοποίηση κάποια στιγμή. Είναι κάτι το οποίο νομίζω θα μπορούσαμε, τουλάχιστον έστω για ένα κομμάτι του τομέα των μεταφορών, να αξιοποιηθεί αυτή η λύση των βιοκαυσίμων από φύκια. Κυρία Σμίτ, ευχαριστώ πολύ και ευχαριστώ θερμά για την παρουσίαση της μελέτης σας. δεν είμαι τόσο θετικά διακειμένη όσο οι προλαλήσαντες. Αν βάλουμε όσο έτος αναφορά στο 2010 με, 20, με μέχρι το 2020 αύξηση κατά 6% της κρίσης των ε, ε, της μείωσης μάλλον των ε, εκπομπών του του, του άνθρακα ή γενικά αερίων του θερμοκηπίου ε, από τον τομέα των μεταφορών πρέπει αντίστοιχα να αυξηθεί σημαντικά η γενικα αεριων του θερμοκηπιου απο τον τομεα των βιοκαυσίμων στις μεταφορές. Ερωτώ λοιπόν, γιατί βλέπω ότι από την έκθεσή σας δεν εκπληρώνουν τα προσδοκόμενα αποτελέσματα τα βιοκαύσιμα. Η χρήση των βιοκαυσίμων θα μπορούσε να οδηγήσει σε αύξηση των ε, αέριων του θερμοκηπίου. Αυτό προκύπτει. Και ένα άλλο πρόβλημα που αναφέρεται επίσης είναι ότι λόγω της αυξανόμενης ζήτησης σε βιοκαύσιμα μειώνεται ή μάλλον αντίστοιχα αυξάνεται η πίεση προς τη χρήση αρρώσιμων ε, εκτάσεων και άρα μπορεί η παραγωγή τροφίμων να δει αρνητικές συνέπειες. Η ερώτησή μου είναι Είναι λογικό όταν έχουμε τόσο περιορισμένους πόρους για την ε, κατασκευή εργοστασίων, αξιοποίηση της ερευνητικής, του ερευνητικού δυναμικού κτλ. Να τους ρίξουμε όλους αυτούς στα βιοκαύσιμα. Μήπως πρέπει να κοιτάξουμε την ηλεκτροκινητικότητα και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας καλύτερα. Να προτιμήσουμε αυτές τις μορφές. Δηλαδή. Ο πρόεδρος ευχαριστώ, θα μιλήσω και εγώ τελευταίος, για τη δεύτερη γενιά. Εάν αξιοποιηθεί αυτή, νομίζω ότι θα καταφέρουμε να αξιοποιήσουμε και τα απόβλητα. Ε, η δεύτερη γενιά όμως πώς μπορεί να εξασφαλιστεί αν δεν έχει ε, λειτουργήσει ικανοποιητικά η πρώτη. Το 20% των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα ξέρουμε ότι προκύπτει από την αποψήλωση των δασών και δεν γνωρίζω κανένα πολιτικό ο οποίο να λέει ότι θα πρέπει. των ε, τροπικών δασών. Δεν ξέρω κανένα πολιτικό ο οποίο να λέει α θέλουμε να καταστρέψουμε όλα τα ε, τροπικά δάση, αλλά Ξέρουμε ότι εκεί μπορεί να έχουν πολύ καλύτερη παραγωγή για τα βιοκαύσιμα. Επομένω, η τάση για παραγωγή βιοκαυσίμων είναι να αξιοποιούνται αυτέ οι περιοχέ των τροπικών δασών. Είναι κάτι το οποίο βλέπουμε σαν ε, προβολή στο μέλλον, δηλαδή ο παραγωγός, ο γεωργικός παραγωγός του εχθές ή του παρελθόντος είναι ο παραγωγός βιοκαυσίμων του μέλλοντος. Αντίστοιχα χρησιμοποιούνται οι ε, αρρώσμες εκτάσεις. Ε, μην φτάσουμε δηλαδή να μην έχουμε αρκετά τρόφιμα και να λιμοκτονούν ε, οι πολίτες επειδή προτιμήσαμε να φτιάχνουμε βιοκαύσιμα. Γι' αυτό νομίζω ότι θα πρέπει να στραφούμε πιο πολύ στην ηλιακή ενέργεια, στην αιωλική ενέργεια. Η Φινλανδία και η Σουηδία έχουν πολλές ακτές, έχουν πολλούς ανέμους. Αν αξιοποιούσαν και μάλιστα μπορούν ολόκληρο το χρόνο να αξιοποιούν την αιωλική ενέργεια. Δεν πρέπει να δούμε αν αυτό είναι πολύ πιο οικονομικό ενδεχομένω από τα βιοκαύσιμα. Ένα άλλο ζήτημα που θα ήταν η επέκταση της υποχρεωτικής της ταχύτητας κατά 30, στα 30 χιλιόμετρα στο ιστορικό των πόλεων παντού. Αυτό θα εξοικονομούσε κατά 12% σε κάψιμα που χρησιμοποιούνται τεράστια οικονομία. Το ίδιο θα μπορούσαμε να δούμε βιοκαύσιμα όπως αυτά που αναφέρατε εσείς για τα φύκια, σαν δυνατότητα έρευνας. Αλλά έχουμε άμεσα τη δυνατότητα να μειώσουμε σοβαρά τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα αν επιβάλαμε τέτοια μέτρα απλά όπως το νατοτόριο ταχύτητα στα 30 χιλιόμετρα ε, και πάρα πολύ γρήγορα. Αυτά λοιπόν τα σχόλιά σας και έχετε το λόγο. Θα προσπαθήσω να απαντήσω σε όλους σας. Για τα όσα αναφέρατε, τα οποία αλληλοσχετίζονται. Οπότε δεν θα απαντήσω χωριστά. Πάντως, το κεντρικό σημείο είναι το πώς τώρα θα αναπτύξουμε τεχνολογία σχετική με τις μεταφορές. Άρα, πέραν του βιοκαυσίου, το θέμα είναι πώς θα έχουμε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας για τις μεταφορές. Είναι προτεραιότητα αυτό το να υπάρχει ένα τοπικό σύστημα ε, μεταφορών. Και εμείς έχουμε δεσμευθεί να δούμε τι διαφορετικές λύσεις μπορεί να υπάρξουν τόσο ώστε να είμαστε όσο είναι πιο αποφασιστικοί. Τμήμα της λύσης είναι τα δύο καύσιμα και όπως ήδη αναφέρθηκε θα πρέπει να εντοπιστεί το πώς η δεύτερη γενναία καυσίμου μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην αγορά πιο αποτελεσματικά. Αλλά όπως ξεκαθαρίσαμε η θέσπιση των δύο ε, αποτελεί τη λύση σε περισσότερα από ένα προβλήματα. Το περιβάλλον, ήδη το είπαμε. Ε, το θέμα της βιωσιμότητας, πολύ σημαντικό. Για τη βιομάζα, για τις ε, ζωοτροφές, για τα ε, υπολείμματα. Επομένως, η βιωσιμότητα σχέση με το περιβάλλον πολύ σημαντικό. Κάτι άλλο επίσης είναι ο παράγον κόστος. Οπότε θα πρέπει να εντοπίσουμε, θα πρέπει να αναπτύξουμε όλα και καλύτερη τεχνολογία για να γίνουμε ανταγωνιστικοί. Και για να γίνουμε ανταγωνιστικοί θα πρέπει να επενδύσουμε στην ε, ανάπτυξη τεχνολογία, στην έρευνα, αλλά επίσης και στην επιστημονική επίδειξη. Προς το παρόν έχουμε πάρα πολύ λίγες εγκαταστάσεις στην Ευρώπη που μπορούν να επιδείξουν σε μεγάλη κλίμακα την βιωσιμότητα των καυσίμων δεύτερη Γενία, άρα πρέπει να επενδύσουμε περισσότερο. Αλλά προ τούτο χρειαζόμαστε πιο μακρόπνο, πιο εξωτερικέ ε, πολιτικό πλαίσιο, γιατί χρειάζεται δέσμευση στα κράτη-μέλη όσον αφορά του χρήστε των καυσίμων δεύτερη Γενιά, επομένω είναι θέμα περιφυβαλλοντικό, είναι οικονομικό, είναι και πολιτικό, όπως βλέπουμε το θέμα του μέλλοντος των δύο Αλλά έχουμε και την τρίτη γενιά η οποία απέχει ακόμη περισσότερο από την ε, πραγματικότητα. Οπότε χρειάζονται εδώ βελτιώσεις ε, παντού. Όπως ήδη είπαμε, σε 10 χρόνια θα έχουμε αυτή την ε, νέα γενιά, η πρώτη γενιά πάντως των βιοκαυσίμων. θα βοηθήσει την τεχνολογία για τις τοπικές μεταφορές, αλλά δεν θα είναι αυτή η μόνη ε, ωφέλεια. Και η κινητικότητα επίσης θα ωφεληθεί από αυτήν την ανάπτυξη νέας τεχνολογίας της μεταφορές. Επίσης, αυτή η κινητικότητα είναι κάτι σαν επανάσταση. Μιλάμε για ηλεκτρική κινητικότητα. Άρα χρειαζόμαστε κάποια οχήματα, σύστημα, ένα ευφύε σύστημα που να το αναπτύξουμε. Δεν είναι ότι φορτίζουμε το όχημα και κατόπιν πάει κάποιος το παίρνει το όχημα. Θα πρέπει στην κατάλληλη τιμή, με την αρίστη τιμή, την πιο συμφέρουσα, έτσι να προσφέρεται ο ηλεκτρισμό. Άρα χρειάζεται τέτοιου είδους ευφύες σύστημα ασφάλεια, προμήθειας, ε, ασφάλεια ενημέρωσης και επίσης ε, αποθήκευση της ηλεκτρικής ενέργειας. Επομένως με το νέο σύστημα θα έχουμε αυτά τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, ηλεκτρικά οχήματα και θα έχουμε την ηλεκτρονική, ηλεκτρική κινητικότητα, πολύ σημαντική για την Ευρώπη. Και είδατε το, το Ίδρυμά μας προσπαθεί να βοηθήσει την ανάπτυξη αυτής της τεχνολογίας και ξεκινάμε τον Οκτώβριο φέτος με τα εγγένεια ενός νέου κέντρου που θα ονομάζεται ε, Κέντρο Διαλειτουργικότητας που θα είναι ακριβώς το ίδιο όπως έγινε και στις Ηνωμένες Πολιτείες προδιετίας ένα εργαστήριο και όλα αυτά θα τα δούμε εκεί πέρα όλα όσα χρειάζεται ως μεταβλητές, ως συστατικά ούτως αυτό το ηλεκτρικό σύστημα πως θα είναι η άδραση; πως τα καινούργια δίκτυα θα μπορούν να εξυπηρετήσουν ε, όλη αυτή την κατανάλωση αλλά και την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας που προέρχεται από αυτά τα οχήματα. Πώς θα γίνει η αποθήκευση της ηλεκτρικής ενέργειας. Ένα νέο σύστημα μεταφορών. Περίπλοκο. Οπότε και τώρα αυτό είναι κομμάτι του θεματολογίου μας. Είναι προτεραιότητά μας. Και η βιοενέργεια είναι τμήμα της λύσης. Δεν είναι η μόνη λύση. Ε, υγρά αέριο, ε, φυσικό αέριο, Υπάρχουν και άλλα καύσιμα. Πολλές παράμετροι θα πρέπει να ληφθούν υπόψη. Και όπω αναφέραμε έχουμε και την βιωσιμότητα. Αναφέρθηκαν τα δάση. Είναι σαφής κατάσταση ότι θα πρέπει τα κριτήρια της βιωσιμότητας να τα σεβαστεί δεύτερη γενιά καυσίμων. Και βέβαια τα θέματα μετά τα διατροφικά, αλλά και το πρόβλημα των δασών. Οι συνεργάτες του παρουσιαστή. Ο κύριος Διευθυντής σας απάντησε σε όλα. Α, να σας πω για τα δάση. Μια που πολλοί συνάδελφοι ανέφεραν τους πόρους α, σχετικούς με τα δάση της Βορείου Ευρώπης. Πολύ σημαντικό για τα βιοκάσιμα και τη βιοενέργεια. Πάντως θα πρέπει να κινητοποιήσουμε αυτούς τους πόρους, να καταβάλουμε τη μεγάλη προσπάθεια που χρειάζεται και με μεγάλη προσοχή να δούμε τι θα πρέπει να ενεργοποιήσουμε, πώς θα γίνει αυτού του είδους η ε, σορευτική χρήση. Είδαμε τι γίνεται με τον χαρτοπολτό, με το χαρτί, με τις ε, οικοδομές. όσον αφορά την χρήση της ξυλίας των δασών και τα υπολείμματα μια που δεν ωφελούν όλα, γιατί υπάρχουν εδώ ζητήματα επιπτώσεων στο περιβάλλον και στο φαινόμενο θερμοκηπείο. Η Φιλανδία και η Σουηδία κάνουν μεγάλη προσπάθεια σε αυτό το μέτωπο. η Φιλανδία είναι η μόνη ευρωπαϊκή χώρα που έχει εγκαταστάσεις ε, παραγωγής διζελ δεύτερης γενιάς. Πουθενά άλλο δεν υπάρχει κάτι τέτοιο στην Ευρώπη. Όπως είπαμε το πρόβλημα είναι το τι κανείς θα κινητοποιήσει. Υπάρχουν ε, πολλά κατάλοιπα των φυσικών πόρων. Αλλά το θέμα είναι το ότι θα πρέπει κανείς να χτίσει, να φτιάξει τις καταστάσεις και να πετύχει ανταγωνιστική τιμή. Δεύτερη γενιά επομένω. Να υπάρξει έρευνα και ανάπτυξη σε τουλάχιστον κλίμακα πριν τη φάση της ε, θέσης εμπορία. Άρα ακόμα υπάρχει πολλοί δρόμος που έχουμε να κάνουμε. Ο Πρόεδρος. Και πότε θα έχουμε την τρίτη γενιά λέτε, ρωτάει η βουλευτής. Α, λέτε για τα κυφίκια. Εδώ η προβλέψη είναι μάλλον πιο αισιόδοξη από την πραγματικότητα, γιατί πραγματικά έχουμε καθυστερήσει πολύ και μόνο έρευνα και ανάπτυξη σε εργαστήρια. Και υπάρχει πιο πολύ ένταση παραγωγής ε, όσον αφορά το θέμα του φαινοκηπίου από ότι οι προηγούμενες γενιές. Και έχουμε τα λιπίδια, τα, τα, και τα άλλα λιπογόνα, ε, ε, οξέα τα οποία παράγονται και άρα έχουμε ε, αυτό είναι αρνητικό, έχουμε μεγάλο κόστος παραγωγής, άρα θα πρέπει να συνδυαστεί η παραγωγή με άλλα υλικά που θα τίθενται σε εμπορία, με άλλου είδους καύσιμα, το οποίο έτσι θα είναι συμφέρον. Όμως υπάρχουν πολλά προβλήματα να επιληθούν πριν από εκείνη τη φάση. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσίασή σας, για τις απαντήσεις. Οπότε εδώ ολοκληρώνεται αυτό το σημείο τη διάταξη και σα ευχαριστώ πολύ, λέει ο Πρόεδρο, για αυτή τη μελέτη, η οποία είναι διαθέσιμη όποιον θέλει. Υπάρχει στα αγγλικά, φαντάζομαι όλοι έχετε λάβει ένα αντίγραφο. Καλησπέρα σα. Η μία έκπληξη διαδέχεται την άλλη. Βλέπω φωτογραφία με καλά, με χρόνια πολλά, με συγχωρείτε. Είναι υπέροχο να δουλεύει κανείς τη μέρα που έχει τα γενέθλιά του με όλες τι ευχέ. Δεν ξέρω πού το μάθατε ότι έχω τα γενέθλιά μου. Η συνάδελφος εδώ είναι πολύ γνωστή, ήταν ευρωβουλευτής όταν ε, ήρθα εγώ το 2004, ήταν υπουργό στην Ολλανδία. Γνωριζόμαστε εδώ και πάρα πολλά χρόνια με την κυρία Πέις και τώρα είναι συντονίστρια για το διάδρομο Ρήνου Δούναβη και με μεγάλη χαρά θα σας ακούσουμε. Σας καλωσορίζουμε λοιπόν και πάλι. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Αξιότιμα μέλη του Κοινοβουλίου. Και αγαπητοί προσκεκλημένοι, σίγουρα πολλές φορές άκουσες πως το πρόγραμμα εργασίας κάθε συντονιστή έχει περάσει από πολλά βήματα διαβούλευσης. Ναι, τέσσερα κάναμε εμείς από τον Απρίλιο του 2004 μέχρι τον Νοέμβριο του 2004 με εκπροσώπους από τα Εθνικά Υπουργεία Συγκοινωνιών, από τις περιφέρειες, από τις τοπικές αρχές, ε, μάνετζερ, ε, αεροπλοεία, εσωτερική ναυσιπλοεία, οδικοί άξονες, τέρμινα λοδικά, σιδηροδρομικά. Όπως ακούσατε κι εσείς για πρώτη φορά έχουμε και τώρα πάω στην περιγραφή του διαδρόμου, κάτι το οποίο καλύπτει μια τεράστια περιοχή και πολύ κοντά στην καρδιά του προέδρου σας, μια και μιλάμε για το Δούναβι, ε, μοιράζεται σε δύο κλαδιά ο διάδρομος αυτός, βορρά και νότο. Το βόρειο κομμάτι είναι η Τσεχία-Σλοβακία στο βορρά και έχουμε στο νότο αυτό του Εύξενου πόντου της Μαύρης Θάλασσας. Εκεί έχουμε δύο διαφορετικές διαδρομές, είναι οδική και σιδηροδρομική. Στο βορρά πάμε Νιρεμβέρκη, Φρακφούρτη και προς το νότο στο Στουτγάρδι, Μόναχο, σαλτσβουργκ Στη Ρουμανία η διαδρομή πηγαίνει στο Σέβες και περνάει και από το Κράγιοβα για τις εσωτερικές, ε, για την εσωτερική ε, ναυσιπλοεία περνάει από το Ρήνο και μέχρι τη Μαύρη Θάλασσα στις εκβολές του Δούναβη. Επίσης από τον ε, Σέμα και φτάνει στο λιμάνι του Σίσακα. Αν εξετάσετε λοιπόν την απόσταση αυτής της πλωτής διαδρομής θα εκπλαγείτε. Ο Δούναβης μόνος του είναι 3.000 χιλιόμετρα περίπου μακρύς. Το κομμάτι στην Τσεχία έχει δύο σημεία αφετηρίας. Έχουμε Πίλσεν και Πράγα μέχρι το Πυρόφ στην Τσεχική Δημοκρατία και μετά Αυτά ξεκινάνε από την Ιρεμβέρια και την Φραγκφούρτη και αν δεν τα προφέρω καλά συγχωρέστε με. Μετά το Πρέροφ και το Γκράνιτσε και τη Μοράβια, σιδηροδρομική αξιγραμμή περνά από την Οστράβα για τους επιβάτες και μία γραμμή από τη Σελίνα και το Πάτσεφ από τη Σλοβακία για τα εμπορικά τρένα όχι βέβαια αποκλειστικά, για την οδική διαδρομή Στρασβούργου, Φραγκφούρτη, Νίρεμβέργη, Πράγα, Μπρουνό, Κόσιτσε, Τσιλίνα και φτάνουμε και στα σύνορα με την Ουκρανία. Για να σας δείξω πόσα κράτη μάλλη εμπλέκονται, να σας πω πως η διαδρομή συνδέει 8 κράτη-μέλη και 4 μη μέλη Σερβία, Βοσνία, Ζεγογίνη, Μολδαβία και Ουκρανία. Και μιλάμε μόνο για τις πλωτές οδούς εσωτερικής ναυσιπλοΐας. Πάνω από 3.500 χιλιόμετρα ε, συντηροδρομικής τροχιάς, 2.700 ε, χιλιόμετρα ε, ποταμών και 7 περίπου χιλιάδες χιλιόμετρα δρόμων πάνω από 30 ε, σιδηροδρομικοί σταθμοί και εσωτερικά λιμάνια, 21 συνοριακά περάσματα. Πολύ σημαντικό αυτό για την Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί αυτό αποτελεί προτεραιότητα, γιατί οι υποδομές σε διασυνοριακό επίπεδο είναι πάντα κάτι το δύσκολο. 8 σιδηροδρομικά, 7 ε, οδικά και 6 ε, πλωτά τέτοια διασυνοριακά περάσματα. 19 κομβικά λιμάνια που είναι πολύ σημαντικό γιατί βέβαια εκεί πρέπει να περνάει ένα συγκεκριμένος όγκος τον κάθε χρόνο για να θεωρήσει κομβικό λιμάνι και 11 αεροδρόμια. Ποια είναι τα κρίσιμα θέματα. Είναι αρκετά περίπλοκο γιατί έχει να κάνει με τη σχέση μεταξύ χωρών που έχουν από τότε που θυμούνται χρησιμοποιήσει τα δικά τους σιδηροδρομικά δίκτυα που συνέδεαν την πρωτεύουσα με την επαρχία και τώρα πρέπει να δημιουργήσουν ένα ευρωπαϊκό διάδρομο για μεγάλες ροές επιβατών και εμπορευμάτων βασιζόμενοι σε τρεις βασικές παραδοχές. Μην ξεχνάτε πως επειδή ακριβώς πρόκειται για ευρωπαϊκό διάδρομο ο Ευρωπαίος φορολογούμενος έχει τη διάθεση να αναλάβει το κόστος. Εάν τα κράτη-μέλη επιθυμούν αποκλειστικά και μόνο να αναλάβουν αυτά που τα αφορούν, τότε πολλά, πολύ λίγα, πολύ λίγους λόγους θα έχει ο Ευρωπαίος φορολογούμενος για να καταβάλει το αντίμητιμο για την δημιουργία αυτών των υποδομών ο Ευρωπαίος φορολογούμενος απερίφραστα δήλωσε πως ναι, αλλά να είναι πραγματικά ευρωπαϊκό σχέδιο. Να είναι ευρωπαϊκής διάστασης αυτή η διάδρομη. Τι είναι σημαντικό λοιπόν. Τρεις παραδοχές όπως σας είπα. Η διαλειτουργικότητα καταρχήν για βιώσιμη και αποδοτικότητα ...για σύνδεση όλων των μέσων μεταφοράς. Υψηλό ποιοτικό επίπεδο υποδομών, για παράδειγμα, υψηλής ε, ταχύτητας ε, τρένα και διαχείριση δικτύου, ε, ελάχιστο φορτίο για τα τρένα, 365 μέρες χρήση των πλωτών δυνατοτήτων και σύνδεση με το οδικό δίκτυο. Αυτά λοιπόν θα πρέπει να είναι τα ίδια παντού. Διαλειτουργικότητα. Και κυρίως στην περίπτωση του σιδηροδρομικού δακτύου που έχουν διαφορετικά συστήματα ηλεκτροκίνησης και πολλές φορές τμήματα που δεν είναι ηλεκτροκινούμενα, όπως επίσης και διαφορετική σηματοδότηση, είναι σημαντικό για την ασφάλεια και για να είναι δυνατόν να είναι πραγματικός σιδηροδρομικός διάδρομος. Άρα λοιπόν θα πρέπει και εκεί να εξασφαλίσουμε πως υπάρχει ευρωπαϊκή διαχείριση σιδηροδρομικών δικτύων και στη σηματοδότηση και στην ηλεκτροκίνηση. Διαφορετικά δεν μπορεί κανείς ε, με, την ίδια, με τον ίδιο σειρμό να ταξιδέψει από άκρη σε άκρη στην Ευρώπη. Επενδυτικά λοιπόν, τι απαιτείται. Μεγάλα ποσά η έκταση του διαδρόμου και οι απαραίτητες επενδύσεις για να εφαρμοστεί σε ψηλά επίπεδα όπως έχουμε δηλώσει οδηγούν σε ένα υπολογιζόμενο κόστος πάνω από 64 δις ευρώ. Αυτό το 64,64 είναι 64 δις 640 εκατομμύρια ευρώ. Τεράστιο. Δύο τρίτα αυτών των κονδυλίων έχουν να κάνουν με την κατασκευή των υποδομών, την αναβάθμιση, τον χρονισμό, όπως επίσης και την τυποποίηση για το Ευρωπαϊκό Σύστημα Διαχείρισης. Ένα τέταρτο ε, σχετίζεται με τους δρόμους που θα χρειαστούν και το 6% θα πάει στους πλωτές ε, ε, διαδρομές. Εκπλήσαμε, λέει ο Πρόεδρος. Αυτό το κάνω για να σας ε, καθησυχάσουμε. Και τέλος είναι η τερματική σταθμή, ε, logistics και πρόσβαση σε αεροδρόμια. Προτεραιότητες λοιπόν. Αν η επιθυμία μας είναι να επενδύσουμε σε διαδρόμους και επαναλαμβάνω, αν κοιτάξετε την έκταση και το μέγεθος του διαδρόμου, όλους ο Ρήνος, όλους ο Δούναβης και ο ποταμός Μάιν, τότε θα πρέπει να θέσουμε προτεραιότητες γιατί δεν μπορούν να γίνουν όλα παράλληλα. Άρα λοιπόν... It's money. It becomes Τότε είναι απαραίτητο να ορίσουμε τις προτεραιότητες τη στιγμή που θα επενδύσουμε γιατί πολλές φορές στα σύνορα έχουμε σημεία συμφόρησης, γιατί τεχνικά μπορεί να έχουν διαφορετικά συστήματα διάφορες χώρες. Αυτό και στο σιδηρόδρομο και στην εσωτερική ναυσιπλοεία. Υπάρχουν αυτά τα εμπόδια έτσι ώστε να υπάρχει ένα κερδοφόρο και βιώσιμο σύστημα. Θυμόσαστε την περίπτωση της Ισπανίας Και βεβαίω τι γίνεται με την περίπτωση της Ρωσίας που δεν είναι βέβαια στην Ευρωπαϊκή Ένωση που έχει διαφορετικό πλάτο τροχιάς. Και βέβαια το θέμα της σηματοδότηση που προκύπτει παντού. Για το Δούναβι να σας πω πως έχουμε ε, συντονισμό των προσπαθειών που κάνουν, γίνονται για την συντήρηση ενός βιώσιμου πλωτού διαδρόμου και εδώ έχουμε ένα master plan για τη διατήρηση που ε, υπογράφηκε από όλα τα παραποτάμια κράτη, είτε είναι μέλη είτε όχι. Πέρσι η Βουλγαρία και η Ρουμανία υπέγραψαν ένα μνημόνιο αμοιβαία συνεργασίας ε, για επίγουσες περιπτώσεις στο κομμάτι του Δούναβη που μοιράζονται. Ξέρετε πως η Ρουμανία και η Βουλγαρία έχουν ένα μεγάλο κομμάτι του Δούναβη και πρέπει να συνεργαστούν έτσι ώστε τα πράγματα εκεί να επιταχυνθούν. Και θα πρέπει βέβαια μαζί να διατηρούν σε καλή κατάσταση το ποτάμι αυτό. Ξέρουμε πως ο δρόμος μπροστά μας είναι μακρύς. Αν δείτε όμως τα έργα τα οποία ανήκουν ε, στο διάδρομο θα δείτε ότι πρέπει να είμαστε έτοιμοι μέχρι το 2030. Εσύ ζητάς κάτι άλλο? Α, μάλιστα. Θα θέλεις το τρένο να κουβαλάει ε, το πλωτό μέσο αντίθετα με το ότι έχουμε στη διαφάνεια μάλιστα. Εν πάση περιπτώσει αυτό είναι το πρώτο σχέδιο το πρώτο σχέδιο ε, προγράμματος εργασίας και νομίζω θα μας βοηθήσει να κατανοήσουμε καλύτερα το θέμα. Και πριν ετοιμάσουμε αυτό το σχέδιο, δεν είχαμε ιδέα για το τι πρέπει να κάνουμε στην Ευρώπη. Και το τι θα πρέπει να συμπεριλάβουμε και πόσο σημαντικές ήταν οι διαφορές. Στόχος μας είναι κάθε χώρα να έχει ένα δίκτυο μεταφορών που χρησιμοποιεί και δρέπει τα πλεονεκτήματα των περιφερειακών του ιδιαιτεροτήτων, δημιουργώντας γέφυρες που θα ξεπερνάνε τα εθνικά σύνορα για σταθερή, βιώσιμη ανάπτυξη στην περιοχή που θα προσφέρει πλέον σε όσους ζουν στις χώρες αυτές και παράλληλα θα διατηρήσει την εθνική κληρονομιά. Κάτι πολύ θετικό, γιατί υπάρχουν υπέροχα τοπία και δεν θέλουμε να τα καταστρέψουμε. Σας ευχαριστώ πολύ. Με χαρά θα απαντήσω σε οποιαδήποτε ερώτηση για το σχέδιο εργασίας και για τις μελλοντικές εξελίξεις στην υπέροχη αυτή διαδρομή Ρήνου Δούναβη. Ευχαριστώ πολύ για την παρουσίαση. Ο Βιμ Φανανκάμπ πρώτος. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Πάντα με μεγάλη χαρά συναντώ και ξανασυναντώ την κυρία Κάρλα Πέις. Είμαστε της παλιάς φρουράς εμείς. Είμαστε το πραγματικό, το γνήσιο ΣΕΝΤΕΑ. Έχω λοιπόν τις εξής ερωτήσεις. Από την Κεντρική Επιτροπή του Ρήνου έχουμε ήδη μια σειρά ε, νομοθετημάτων. Μπορούμε αυτά να τα αξιοποιήσουμε για τον Δούναβη. Μπορεί να γίνει μια προσαρμογή ταχεία. Γιατί νομίζω ότι αξίζει τον κόπο. Δεύτερον, οι επενδύσει της Κίνας. Υπάρχουν θετικές, υπάρχουν αρνητικές Ε, συνέπειες. Μπορούμε να αξιοποιήσουμε αυτό, ε, αυτές τις επενδύσεις τις κινέζικες, κυρίως στη γραμμή της Βουδαπέστης και του Βουκουρεστίου. Έχει επίσης η ρουμανική κυβέρνηση αποφασίσει να κλείσει μια σειρά από γραμμές συντηροδρομικές. Αυτό επηρεάζει τις δικές σας ε, εργασίες, τη δουλειά που κάνετε για τον διάδρομο. Και μια ακόμη ερώτηση που αφορά το μέλλον. Ε, και που έχει σχέση με τον Έλβα ποταμό. Θα μπορούσε ο Έλβας να συνδυαστεί με το Δούναβι στο μέλλον. Παρακαλώ, επόμενος ομιλητής. Χθες είδαμε τον απολογισμό της Λετωνικής Προεδρίας ε, και είπαν πολλοί συνάδελφοι ότι είναι πάρα πολύ σημαντική η διάσταση των εσωτερικών πλωτών οδών. Θα θέλαμε όλοι ο Δούναβης να μετατραπεί σε ένα πραγματικό πλωτό ποταμό. Η φύση τον έχει πρικίσει με όλα τα πλεονεκτήματα. Το πρόβλημα είναι μόνο ότι, και το, είπαν και στον, το είπε και στον ότι υπάρχουν κάποια σημεία ε, όπου δεν, λειτουργεί, δεν μπορεί να λειτουργήσει ως πλωτή οδός, υπάρχουν δηλαδή κάποιες στενοποί και όπου θα πρέπει να εξασφαλιστεί μια διαλειτουργικότητα ενδεχομένω με τις σιδηροδρομικές μεταφορές. Και αυτό αφορά το μέσο και το κατώτερο τμήμα του Δούναβη. Φυσικά πρόκειται για μια μεγάλη πρόκληση. Το είδαμε άλλωστε και στην παρουσίαση με το χάρτη το δίκτυο των ε, οδών και των σιδηροδρόμων ακολουθούν μία γραμμή κατακόρυφη. Δεν υπάρχουν ουσιαστικά οριζόντιες δηλαδή ε, γραμμές που να τέμνουν το Δούναβι. Αυτό θα χρειαστεί να ε, κατασκευαστεί. Και βέβαια δεν αναφέρομαι μόνο σε δρόμους και σιδηροδρόμους. Θα χρειαστεί να αναπτυχθούν και περιφερειακά ε, περιφερειακοί ποταμοί όπως η Τσίσε, όπως ο Σάβα, Κροατία, Σλοβακία, Ουγγαρία, Ρουμανία πρέπει να συνδυαστούν. Πρόκειται για ποταμούς σημαντικούς για τις χώρες αυτές και ίσως έτσι μπορούμε να συνδέσουμε με διάφορες περιοχές τον Δούναβε Και βέβαια δεν ανέφερα και, το, και τη Σερβία, όπου επίσης θα χρειαζόταν πολύ υποστήριξη και επενδύσεις. όπως είπε και ο συνάδελφος Φαντανκάμπ, υπάρχουν ε, κινέζικες επενδύσεις. Και Άραβες ε, επίσης ενδιαφέρονται για επενδύσεις τους στον τομέα αυτών τα επόμενα χρόνια. Γι' αυτό νομίζω ότι πρέπει ο Δούναβης να ενσωματωθεί στην οικονομία μας και στο κομμάτι αυτό της Ευρώπης που είναι και η δική μου πατρίδα η Ουγγαρία αλλά και γενικά η Κεντρική Ανατολική Ευρώπη χρειάζεται ένα δίκτυο οριζόντιας από Ανατολάς προς Δυσμάς δηλαδή κατεύθυνση. Και διασύνδεση του Ρούβου του Δούναβη με τις ε, γειτονικές και μικρότερες πλωτές οδούς που μπορεί να φαίνεται περιφερειακό έργο αλλά έχει μεγάλες ε, διαστάσεις και δυνατότητες. Πρέπει να υποστηρίξουμε το Δούναβι ως πρωτή οδό και να τον ενσωματώσουμε πλήρως στην οικονομική μας δραστηριότητα. Θα ήθελα να ακούσω τη γνώμη της ε, συντονίστριας. Ευχαριστώ Μαρινέσκου. Thank you, uh, Chair. I have three questions. Έχω τρεις ερωτήσεις κύριε Πρόεδρε. Κατά αυτή την περίοδο τα κράτη-μέλη εκπονούν αυτό το μείζον πρόγραμμα. Και σας ερωτώ, Πώ θα φροντίσετε την εναρμόνιση μεταξύ των διαδρόμων. Όχι μόνο για αυτόν, για όλους που καλύπτονται από αυτά τα μείζωνα ε, προγράμματα. Για την περίοδο 14 έως 20. Και έτσι να προχωρήσουμε σε έργα και σχέδια μέσα στους επιμέρους ε, διαδρόμους. Δεύτερη ερώτηση. Ο Δούναβης είναι ένα ποτάμι και αν κράτος δεν κάνει αυτό το οποίο πρέπει, τότε δεν ωφελεί ακόμα και αν όλα τα άλλα κράτη που βρέχονται από το Δούναβι κάνουν αυτό που πρέπει. Άρα πώς θα το φροντίσετε αυτό, γιατί ας πούμε, για παράδειγμα, η Ουγγαρία δεν ενδιαφέρεται και τόσο πολύ στο να επενδύσει ε, ε, για τον Δούναβι. Τρίτον, εσείς τι πρόγραμμα εργασίας έχετε, πέστε μας ξεκάθαρα. Μας είπατε, θα κάνετε το α, το β, το γ. Πώς θα το κάνετε και πότε και με τι χρηματοδότηση, όπου θα βγει αυτή η χρηματοδότηση. Υπάρχει κάποιο πραγματικό ε, πρόγραμμα εργασίας. Η κυρία Μάσινερ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ τη συντονίστρια. Δεν χρειάζεται να ρωτήσω τίποτα για τους συνδεδρόμους της Ρουμανίας. Το κάλυψε ο, ο Ευτυχώ, ε, αλλά θα ήθελα να συναντήσω τον κύριο Μαρινέσκου σε μια ερώτηση, γιατί σήμερα το πρωί η κυρία ε, Τροτμάν αναφέρθηκε σε πέντε πιο σημαντικά σχέδια που αφορούν το διαδρομό της. Εσείς έχετε κάτι αντίστοιχο, αν όχι πέντε έστω και λιγότερα, αλλά πιο σημαντικά ε, σχέδια προτεραιότητας. Και επίσης ακολουθούν οι κυβερνήσεις τις επιλογές τις οποίες έχουμε προβεί εμείς για τα πιο σημαντικά έργα, εκεί δηλαδή που χρειάζεται να κλείσουν κάποια κενά στους ε, διαδρόμους ε, ή ε, έργα που έχουμε πάση περιπτώσει επιλέξει. Υπάρχουν αντίστοιχα προτάσεις για κατασκευές από τις κυβερνήσεις και για τις εσωτερικές πλωτές οδούς, όπως και ο ΒΙΜ είμαι και εγώ ένθερμη υποστηρίκτρα των εσωτερικών πλωτών οδών, η κυρία Τιτσάουρ μας λέει ότι θα πρέπει ο Δούναβης να είναι πάντα ένας τρόπος διασύνδεσης μεταξύ Ατλαντικού και Μαύρης Θάλασσας. Να μπορούν να μεταφέρονται όλα ε, ναυσιπλοϊκώς από τη μια θάλασσα στην άλλη. Εσείς πώς το βλέπετε αυτό. Γιατί δεν νομίζω να υπάρχει κανείς από τον κλάδο των μεταφορών που να το αποκλεί, αλλά ασφαλώ θα πρέπει να καταστεί πλωτό ο Δούναβη σε όλα τα σημεία. Υπάρχει αυτή η δυνατότητα, ανεξαρτήτως των καναλιών που μπορεί να ανοίξουμε των διορίγων, ε, ο Δούναβης ε, θα πρέπει να είναι ολόκληρος πλωτός. Τώρα θα ήθελα και εγώ να λάβω το λόγο, λέει ο Πρόεδρος, δεν θα ξαφνιαστεί η Καρλαπέης. Δύο, δύο ε, κομπλιμέντα καταρχάς, ότι χαίρομαι ιδιαίτερος που μιλούμε για τον Δούναβη ιδιαίτερος ε, και είπε η Κάρλα Πέις ότι είναι σημαντικές οι προτεραιότητες το σημειώνω αυτό με τρία θαυμαστικά διότι βεβαίως εάν θέλουμε να κάνουμε τα πάντα και τον Μάιν και τον Δούναβη και τον Ρίνο, τότε προφανώς θα χρειαστούν 50 χρόνια. Εάν όμω δώσουμε έμφαση και προτεραιότητα στον Δούναβη και πούμε εδώ χρειάζεται να κάνουμε τη διασύνδεση με το συντηρόδρομο, τότε επικεντρωνόμαστε σε αυτό, αναπτύσσουμε την ιστορική αυτή πλωτή οδό του Δούναβη και προχωρούμε. Και βλέπω ότι έχετε κάπου σημειώσει well established. Ξεφνιάζομαι. Γιατί? διότι έχουμε την διασύνδεση από τον Ατλαντικό μέχρι τη Μαύρη Θάλασσα μέσω της διόρυγας Ρήνου, Μάιν, Δον, Δούναβη με κόστος δισεκατομμυρίων. Ε, ξεκίνησε αυτό από ένα, από μια, σε μια περίοδο της ιστορίας. Ο επόμενος υπουργός πράσινος, ε, σώμα, όχι πράσινος, της ε, Γερμανίας είπε «Α, όχι, δεν γίνεται να ε, προχωρήσουμε αυτό το κανάλι» γιατί οι προγνώσεις έλεγαν ότι θα έφτανε το πολύ πολύ σε 10% αξιοποίηση. Δηλαδή δόθηκε τόσο χρήμα σε υποδομές χωρίς να υπάρχει σχετική ανάγκη. Και γιατί δεν υπήρχε ανάγκη, γιατί τα τελευταία 20 χρόνια οι εσωτερικές πλωτές οδοί ε, μειώθηκαν κατά σημαντικό ποσοστό στην Ευρώπη. Από 20% των μεταφορών έφτασαν στο, έπεσαν στο 8%. Γιατί δεν αξιοποιούνταν επαρκώς. Λοιπόν πρέπει να κοιτάξουμε τι θέλουμε να κάνουμε. Είναι πλωτό ο δουναδή. Εγώ έχω περάσει από το Ingolstadt μέχρι τη Μαύρη Θάλασσα με το ποδήλατο παράλληλα στο με το θαλάσσιο ποδήλατο στον Δούναβη, που βέβαια είναι πολύ εύκολο να ανατραπεί και πρέπει να προσέχει κανείς όταν έρχεται ένα μεγαλύτερο σκάφος να το αποφεύγει κτλ. Πριν από τρία χρόνια αντίστροφα, ποδηλατώντας αυτή τη φορά, είδα μόνο τρία μεγάλα πλοία. Ενώ την προηγούμενη, την πρώτη φορά που είχα κάνει τη διαδρομή ε, κατεβαίνοντα ήταν πάρα πολλά αυτά που είχα συναντήσει. Γιατί, γιατί δεν υπάρχει ζήτηση. Γιατί δεν έχουμε επαρκώς established, όπως λέμε, δηλαδή αρκετά ανεπτυγμένε ανεπτυγμένες ε, εσωτερικές ελάσεις ε, πλωτές οδούς. Πρέπει να κοιτάξουμε το Δούναβι. Βεβαίως μπορεί στην, ε, στην έκταση της Γερμανίας, της Αυστρίας να είναι ικανοποιητικά τα αποτελέσματα, αλλά πρέπει να κοιτάξουμε να είναι παντού πλωτός. Και γι' αυτό θέλω να ρωτήσω αν υπάρχει μια νέα αντίληψη του να αξιοποιούμε τους ποταμούς, να είναι πλήρω προσαρμοσμένη στις ανάγκες των σκαφών ή αν αντίστροφα υπάρχει ενδεχομένως και η τάση να προσαρμόσουμε τα σκάφη στην γεωγραφική, στην γεωφυσική εικόνα των ποταμών. Γιατί ίσως εκεί θα μπορέσουμε καλύτερα να τους αξιοποιήσουμε. Αυτή είναι η ερώτησή μου. Αυτό μπαίνει μέσα στον διάδρομο. Υπάρχουν ε, τα ε, σχέδια για τις προτεραιότητες. Με ξαφνιάζει αυτό που λέτε μόνο 6% για τις πρώτες και το λοιπό στους, το, στους σιδηροδρόμους. Περιμένω να ακούσω τις απαντήσεις σας, κυρία Πέης. Mr. Chairman. Κύριε Πρόεδρε. Then you always between us. μεταξύ μας, μεταξύ μας μόνο. Θα αρχίσω από τις ερωτήσεις του Ολλανδού συναδέλφου. Ερώτησε τι γίνεται με τις διατάξεις που διέπουν την πλεύση ε, στον, Δούνα, στον ε, Ρήνα μπορούν αναλογικά να παραμοστούν και στον Δούναβη. Υπάρχει μια επιτροπή αρμόδια για τον ε, Ρήνο και άλλη αρμοδία για τον Δούναβη. Αυτό που θέλουμε είναι να υπάρξει εξυγχρονισμός. Επί χρόνια προσπαθούμε αυτό να το καταφέρουμε. Και ό,τι είναι δυνατόν να εφαρμοστεί αναλογικά να εφαρμοστεί από το ένα ποτάμι στο άλλο. Πάντως, χρειάζεται και είναι και σημαντικό να υπάρξουν σκάφη τα οποία από τον Ρήνο να περνούν στον Δούναβη χωρίς να χρειάζεται να εφαρμόσουν άλλο πλέγμα κανόνων δικαίου. Επομένως αυτό τραπασχίζουμε τον εξυγχρονισμό της νομοθεσίας που είναι αρμοδιότητα της Επιτροπής για τον Δούναβη. Υπάρχουν και πολιτικά θέματα. Πάντως, φυσικά και θέλουμε να επιταχυνθούν οι ρυθμοί των εργασιών, αλλά όπως είπα, φράγμος είναι κάποια πολιτικά ζητήματα. Τώρα, τα κεφάλαια επενδύσεις από την Κίνα που ανέφερε κάποιος συνάδελφος. Ένα είναι βέβαιο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη-μέλη δεν μπορούν να τα χρηματοδοτήσουν όλα. Είδατε τη σχετική διαφάνεια ότι έχουμε τεράστιες οικονομικές ανάγκες. Και εδώ πέρα λέμε μόνο και μόνο για τους διαδρόμους, γιατί υπάρχουν και άλλου είδους διασυνδέσεις των κρατών μελών. Και μέχρι το 2030 δεν μπορούμε να τα έχουμε κλείσει όλα. Αν θέλουν τα κρατημέλη να προσφύγουν σε δανεισμό από Κίνα και από τους Άραβες. Αυτό δεν μπορούμε να το εμποδίσουμε. Αλλά φυσικά υπάρχουν και ανταλλάγματα για αυτά τα δάνεια. Η ρωμανική κυβέρνηση κλείνει τους δρόμους. Συνάντησα και ζήτησε πολύ ενδιαφέρον πράγματα με τον ομολογό μου της ε, ρωμανικής κυβέρνησης. Και εμείς που λέτε, κλείσαμε μεγάλο τμήμα του σιδηροδρομικού δικτύου. Ε, το κάναμε λίγο μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και το μετανιώσαμε πικρά. Αυτό είπα στον ε, Ρωμανό Υπουργό. Σκεφτείτε το ξανά. Ακόμα και αν δεν χρησιμοποιείτε τον σιδηρόδρομο. μην καταργήσετε τα τρένα. Ξανασκεφτείτε το. Και ξανασκεφτείτε το. Γιατί τώρα έχετε σιδόδρομο, αλλά άμα το καταργήσετε δεν θα το ξανά έχετε. Έχετε το χώρο για τις γραμμές και αν χρησιμοποιήσετε κάποιο άλλο χώρος δεν θα τον ξαναβρείτε ποτέ. Και θα το μετανιώσετε πικρά κάποια μέρα. Κατόπιν, η σύνδεση με τον Έλβα. Δεν καλύπτεται από τον διάδρομο για τον οποίο συζητάμε. Αλλά έχουμε διεξαγάγει έρευνα όσον αφορά τη σχετική σύνδεση Έλβα ΕΛΒΑ-ΔΟΥΝΑΒΕ Στη συνεργασία και με τον πρόεδρο της ε, τσεχικής δημοκρατίας. Συγγνώμη, είπα Τσεχοσλοβακία, αλλά τι να κάνουμε, ε, είναι της εποχής μου. Και κατέληξα και πιστεύω ότι εάν θέλει κανείς να κάνει μια σύνδεση με τον δούναμι, δούναβη χρειάζονται εμπορευματικές μεταφορές. Βέβαια δεν υπάρχει σύνδεση Αμβούργο Πράγας με σκάβους, με πλωτή στο Γιατί γνωρίζουμε ότι η Τσεχία έχει ένα νησάκι στο λιμάνι του Αμβούργου. Δεν θα εξευρεθούν αρκετά εμπορεύματα ούτως ώστε να αξίζει να γίνουν σχετικές επενδύσεις που είναι πάρα πολύ μεγάλες. Πρέπει κανείς να κάνει έργα μέσα από βουνά και εγώ δεν ξέρω τι άλλο. Κοστίζει πάρα πολύ, επομένω χρειάζονται εμπορεύματα προς μεταφορά. Αλλιώς δεν μπορεί να αρχίσει αυτό το έργο της ε, διασύνδεσης. Και πρώτα θα γινόταν ε, για να καλυφθούν αυτά τα εμπορεύματα η σύνδεση με το Αμβούργο. Κύριε Ντέλια. Ότι μου είπαν τα σημεία συμφόρηση στην Βουδαπέστη υπάρχουν. Και ότι οι Κινέζοι και Άραβες ασχολούνται με τον Σάβα και με τον Τίσα. Ο Σάβα, ο συγγνώμη, καλύπτεται από τον διάδρομο. Εξετάζουμε και τα δύο πάντως ποταμιά και τον Τίσα και τώρα αφορά τη Σερβία για την οποία ε, μιλήσατε. Είναι ειδική περίπτωση η Σερβία. Διότι όλα τα σημεία συμφόρηση που υπάρχουν την κάνουν από την αρχή καλή διαχείριση. Ασχολούνται πάρα πολλέ μη κυβερνικές οργανώσεις και φιλοπεριβαλλοντικέ. και αυτό είναι σημαντικό γιατί στη Ρουμανία είχαμε πρόβλημα ως προς αυτό. Άρα, θα πρέπει να δούμε πόσα χρήματα χρειάζεται η Σερβία. Αυτό είναι το πρόβλημα, ακόμα δεν ξέρουμε. Αλλά για τη Σερβία προβλέπονται πολλά διασυνοριακά έργα. Άρα μπορεί να υπάρξει χρηματοδότηση από τα κράτη-μέλη αυτά τα έργα καλύπτονται, όπως καλύπτονται και τα σημεία συμφόρησης. Απλώς θα πρέπει να δούμε αν θα αποδεσμευθούν τα απαραίτητα κονδύλια. Μόνο έτσι οριζόντια που να δουλέψουμε. Χρειαζόμαστε ένα δίκτυο. Και εάν σε κάποια χώρα δεν λειτουργούν τα, τα πράγματα, τότε τίποτα. Για το δεν αυτή να σας πω. Κάνουμε κάτι άλλο. Είναι τόσο μεγάλος ο Δούναβης. Να, ξέρετε, έχουμε σωρό κανάλια στην Ολλανδία. Αλλά φτάνουν τα, ξέρω 200-300 χιλιόμετρα, ενώ ο Δούναβης είναι 2.800 χιλιόμετρα. περνάει και από τα νέα κρατημέλια. Μα γι' αυτό νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σπουδαία υπόθεση ο Δούναβης όσον αφορά τις ε, μεταφορές. Και υπάρχει εδώ η παρεξήγηση. Δεν το έχει καταλάβει και ο πρόεδρός σας όσον αφορά το πόσο κανείς πρέπει να ε, επενδύσει σε τρένα και πόσα σε ποτάμια. Φτάνει σε περιοχή που το χρειάζονται το τρένο. Εγώ επί υπουργείας μου ποτέ δεν είδα ένα δρόμο, μια συνδρομική γραμμή που να μην πηγαίνει σε κάποια περιοχή που καλύπτεται από κάποιο έργο. Δηλαδή θα πρέπει κανείς να προσέξει τη φύση, θα πρέπει να ενεργήσει πολύ προσεκτικά. Πρέπει να κατασκευάσετε πολλές συνδρομικές γραμμές Α, όμως τα χρήματα δεν μπορούν να καλύψουν και το σιδόδρομο και τον Δούναβη και να είναι κανείς και πρόχειρος με το περιβάλλον. Πρέπει κανείς να είναι βέβαια και πρακτικός. Έτσι να αντιμετωπίσει κανείς την περίπτωση του Δουνάβη. Uh, uh, uh, Για να δούμε, επί το παρόντος ε, είναι συνεργάσιμη η Ουγγαρία. Κάνουν ό,τι μπορούν τόσο ώστε να θυραμιστούν με τις προσπάθειες των άλλων χωρών. Άρα υπάρχει ελπίδα. Κύριε Μαρινέσκο. Ε, uh, ε, ε, είπατε για το μείζον πρόγραμμα, το μείζον σχέδιο όλων των διαδρόμων. Έχουμε εννέα διαδρόμους ε, σε κάποια μέρη συγκλίνω όπως στη Γερμανία που πρόκειται για έξι διαδρόμους και έχουμε έρθει σε επαφή με την Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση στη Γερμανία σε σχέση για όλους τους διαδρόμους. Ε, για να δούμε πώς θα ρυθμιστεί η διασταύρωση των διαδρόμων, πώς θα ρυθμιστούν όλα αυτά πιο εύταχτα, πιο, πιο καλά. Μέχρι τώρα Πάει καλά η υπόθεση. Αυτό είναι η δουλειά του συντονιστή. Ότι ο διάδρομος είναι πραγματικός διάδρομος. Ότι δεν διακόπτεται, ότι δεν έχει σημεία συμφόρησης. Γιατί αυτό πάνε να πει διάδρομος. Πάντως επί του παρόντος δεν γνωρίζουμε ποια ήταν αποτέλεσμα τη αξιολόγηση για τα έργα και τα σχέδια. Ε, τώρα, τώρα βρίσκεται την εξελίξη η αξιολόγηση και οπότε δεν ξέρουμε επομένω τι θα εγκρίνει. Άρα δεν μπορώ να σα πω τίποτα από το παρόντο. Όμως αυτή είναι η ουσία τη δουλειά μου. Ότι τελικά να υπάρξει αυτό ο διάδρομος, να λάβει αργά και ωστά. Α, για την Ουγγαρία, όπως είπα στον συνάδελφο τον Ούγγρο, η Ουγγαρία συνεργάζεται μια χαρά τώρα. Από πού τώρα θα προκύψουν τα κονδύλια, από τα διευρωπαϊκά δίκτυα. Γι' αυτο τα κεφάλαια, αυτους του πόρου μιλούμε. Τώρα έχουμε έναν διαγωνισμό, που βολει προσφορών, πρόκειται για 12 δις και θα γίνει επιλογή των σχεδίων και έργων τώρα για τη Ρουμανία. Είναι χρήματα των Ευρωπαίων φορολογουμένων. Γι' αυτό και θέλουμε η διάδρομη να είναι όχι εθνική αλλά ευρωπαϊκή. Κύριε κυρία ποιο είναι το top 5, τα πέντε κορυφαία. Θα σας πω τον επόμενο μήνα ή το φθινόπωρο. Δεν γνωρίζω τον. Διότι κάθε έργο τώρα υφίσταται αξιολόγηση. τα αξιολογούμε, τα αναλύουμε. Άλλα τα πάνε καλά, άλλα τα πάνε χειρότερα, αλλά τέλος πάντων θα πρέπει να περιμένουμε τη δεύτερη φάση. Να έχουν ούτως υπήν όριμάσει. Άρα τώρα δεν μπορώ να απαντήσω. Επίσης, το πρόγραμμα εργασίας το έχετε λάβει. Πρόκειται για συνεργασία, συμφωνία με τα κρατη θα επιλεγούν όσα είναι πιο προτιμητέα, πιο αρεστά. Οπότε προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε με το Δούναβι. Δεν νομίζω ότι υπάρχει επικοινωνία με κάποιο σκάφος Ρότερνταμ, Κωνσταντζα. Έχουμε ενδιάμεσα άλλα, ίσως έχουμε Ρότερνταμ, Βιέννη, μια διαδρομή. Τι να σου πω, εγώ ένα καπετάνιος θα πήγαινα γύρω-γύρω. άμα ήθελα να πάω από το Ρόταμ στην Κωνσταντζα. Δεν θα πήγαινα από το ποτάμι. Κύριε Πρόεδρε, κυρία μου, θα πάντα Πρόεδρο. Κύριε Κράμερ, το αναφέρω γιατί αυτό το ρωτήσατε. Ναι. Βεβαίω και πρόκειται να τάξουμε και προτεραιότητε και φυσικά πρόκειται για ε, σημαντική υπόθεση για του Ευρωπαίου που μπορούν να πάρουν ένα τρένο και να ταξιδέψουν με τρένο παντού σε όλη την Ευρώπη. Αυτό μπορείτε να το δείτε στο κείμενό μα ξεκάθαρα. Αλλά όχι με το τρένο μόνο, να μπορούν να χρησιμοποιήσουν και του ε, πλωτέ οδού, ποιο είναι πιο φτηνά από ότι τα τρένα. Γι' αυτό σα λέω ότι αξίζει τον ε, κόπο κάτι να κάνουμε. Επίσης είναι και πιο ασφαλές όταν μιλούμε για ε, μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων. Γιατί είναι θέμα το αν διασχίζει κανείς σε πόλεις, αν διασχίζει κάποιες ευαίσθητες περιοχές. Τι να σου πω, κάπως είναι το θέμα τι, τι προηγήθηκε το αυγό ή η κότα. γιατί όντως χρησιμοποιήθηκε στο παρελθόν πολύ ο Δούναβης. Αλλά πέραν του πότε, πότε υπάρχει η εποχή των βροχών, έχει τόσα πολλά ειζήματα ο Δούναβης που κολλάνε τα καράβια. Να εξογγείλουν. Άρα τώρα δεν είναι κατάλληλη εποχή για να πλέψει, να διαπλέψει κανείς το Πάντως, υπάρχει περιθώριο να γίνουν πολλά. Να κάνουν πολλά με το Δούναβι και παράλληλα να καταφέρουμε να παραμείνει όσο όμορφος είναι και τώρα. Νομίζω απάντησα σε όλες τις ερωτήσεις. Πρόεδρος. Ευχαριστώ πολύ για την παρουσίαση, ευχαριστώ για τις απαντήσεις. Διατηρούμε την επαφή, εάν υπάρχουν ερωτήσεις. Θα, μας, σας στείλουμε επιστολή και θα απαντήσετε φαντάζομαι στην Κεζίνα Μάισνερ για τις πέντε προτεραιότητες σας όταν έρθουν. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, συνεχίζουμε και καλωσορίζω τον Λόρενς Ιαν Μπρίνκχορστ, Ευρωπαίος Συντονιστή, για το Μεσογειακό Διάδρομο. Κύριε Μπριγκχόρστ, έχετε το λόγο. Thank you. Ευχαριστώ. Πρόεδρε, με χαρά ξανάρχομαι στο Κοινοβούλιο και στην Επιτροπή των Μεταφορών για να συζητήσουμε την, ε, τις εξέλιξεις σχέση με το διάδρομο της Μεσογείου. Θα θυμάστε ασφαλώς ότι από τις αρχές του 2014 μπήκαμε σε μια νέα φάση επεκτείνοντας το διάδρομο και υιοθετώντα τις ε, ε, προτάσεις. Δεν θα μπω όμω στα γενικά θέματα που αφορούν τον διάδρομο γιατί έχετε κάνει τη συζήτηση, έχετε την έκθεση των όλων των συντονιστών. Τα επόμενα 10 λεπτά λεπτών λοιπόν που έχω στη θέσή μου θα τα αφιερώσω στον μεσογειακό διάδρομο που, του οποίου έχω και την ευθύνη. Έχετε λάβει το σχέδιο εργασίας, το πρόγραμμα εργασίας. Μελέτη λοιπόν το 2014 για το μεσογειακό διάδρομο που προκύπτει ως ε, παράγωγο της ε, δουλειάς των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής εξωτερικών ε, παραγόντων με προεδρία του υποφαινομένου και με διάφορες, διάφορες σημεία επαφής. Θα δείτε εδώ πέρα ορισμένα από τα χαρακτηριστικά του διαδρόμου. Διατρέχει έξι κράτη-μέλη, τρία στη Δυτική και τρία στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη. Πρόκειται για το βασικό ε, διάδρομο μεταφορών που πάει από Ανατολάς προς ΣΜΑ στα νότια των Άλπαιων. Ξεκινάει από την ε, Ισπανία και φτάνει μέχρι τα, τα Ουκρανικά σύνορα της Ουγγαρίας. Περνάει τη Γαλλία, της Άλπης προς την Ιταλία προς Ανατολάς, δηλαδή Σλοβενία, Ουγγαρία μέχρι τα ανατολικά της σύνορα με την Ουκρανία, όπως είπαμε. Βλέπετε κάποια από τα χαρακτηριστικά του. Και προσθέτω δύο στοιχεία συνολικό μήκος 3.000 χιλιόμετρα. Πολύ ενδιαφέρον δε και υπογραμμίζει νομίζω και την ευρωπαϊκή διάσταση. Τέμνη 7 εκ των λοιπόν διαδρόμων. Έχει λοιπόν σαφή στρατηγική διάσταση και δεν αφορά μόνο, δεν καλύπτει μόνο διμερείς ανάγκες. Εξασφαλίζει διασύνδεση για όλη την Ευρώπη και βέβαια η γεωπολιτική του διάσταση με την εσωτερική αγορά είναι σαφής νομίζω. Σημαντικό επίσης και καταγράφεται στο πρόγραμμα εργασίας είναι ότι καλύπτει τον, το 18% του ευρωπαϊκού πληθυσμού και το 17% του ΑΕΠ της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πιο σημαντικές οικονομικές ε, περιοχές είναι η Λομβαρδία, η ε, Άλπης, Ροδανός, Καταλωνία, Μαδρίτη, Γαλλία, Ιταλία, Ισπανία εν Αλλά όπως είπα, πρόκειται για τον κύριο, μοναδικό κύριο διάδρομο διασύνδεσης των τύριων των Εδώ έχουμε τα κρίσιμα θέματα. Στην επόμενη διαφάνεια χρειάζεται να καλυφθούν κάποια στοιχεία, κάποιες πτυχές κρίσιμης σημασίας για τη βελτίωση των υποδομών, του δυναμικού και της διλειτουργικότητας. Η εμπειρία έχει δείξει και νομίζω θα συμφωνήσουν οι συναλφοί ότι είναι πολύ δύσκολο τα ε, κομμάτια που διασχίζουν σύνορα να κατασκευαστούν όταν υπάρχουν ε, προδιαγραφέ που σημαίνουν ότι θα χρειαστεί συνεργασία μεταξύ κρατών μελών. Ξέρετε, είναι κάτι το αφύσικο να συνεργάζονται τα κράτη-μέλη. Η εθνική διάσταση δηλαδή είναι αυτή η οποία παίρνει το πάνω χέρι και γι' αυτό και η δική μου η δουλειά, όπω και των λοιπόν στον ιστό, είναι πάνω απ' όλα να εστιαζόμαστε σε αυτά τα ζητήματα διασυνοριακά λοιπόν τμήματα που χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή για τον εξυγχρονισμό, αναβάθμιση και τα λειτουργικά ζητήματα. Δύο παραδείγματα. Μεταξύ Ισπανίας και Γαλλίας υπάρχει μια νέα γραμμή υψηλής ταχύτητας, 2013 ξεκίνησε, είναι όμως υπό ε, είναι περιορισμένη εκμετάλλευση γιατί προτιμούν οι σιδηροδρομικές επιχειρήσεις να χρησιμοποιούν τις ιστορικές γραμμές, δηλαδή να σταματάνε στο σύνορο, να ξεφορτώνουν, να ξαναφορτώνουν και να συνεχίσουμε την αντίστοιχη εθνική γραμμή, προκειμένου να μην χρειαστεί να προσαρμοστούν στη διαβάθμιση την ευρωπαϊκή. Το ίδιο και από την Γαλλία στην Ιταλία, όπου υπάρχει μια παλαιά ε, σιδηροδρομική γραμμή, 1870 ε, κατασκευάστηκε, 150 χρόνια πριν δηλαδή, από τη γαλλική πλευρά χρειάζεται διπλούς διπλές μηχανές και περιορίζεται λόγω των διαφόρων γωνιών που έχει αυτή η γραμμή το μήκος του σειρμού. Χρειάζεται οπωσδήποτε κάτι διαφορετικό για να καλυφθεί η γραμμή λιών ζυρίχης. Ε, Επίσης ε, θα πρέπει να δούμε τις ε, ε, την ευθυγράμμιση προδιαγραφές TNT ε, για όλες τις γραμμές, μέσο και μακροπρόθεσμα. Περιορισμοί υπάρχουν σε όλα τα αστικά κέντρα ουσιαστικά, με διαφορετικές λύσεις ε, και περιορισμού σε σχέση με τις δυνατότητες αξιοποίησης των μέσων σταθερής τροχιάς. Ιδιαίτερα στη συνδρομική γραμμή μεταξύ Μομπελιέ και Περπινιά. Όταν αναπτυχθούν όλες τι συνδέσεις με μεταξύ των περιοχών αυτών και των ισπανικών ε, λιμένων, θα φτάσει στα ωριά του το σύστημα. Η νέα γραμμή θα καταστεί δυνατή λοιπόν και ε, απαραίτητη και για να αξιοποιηθεί το πλήρες δυναμικό του διαδρόμου. Μέχρι το 2030, 15 χρόνια δηλαδή μετά, θα χρειάζεται ίσω και 300 τρένα την ημέρα η γραμμή του Μομπελιέ, 140 φορτηγά τρένα 130 περιφερειακά και πολυάριθμα ταχείας, ε, υψηλής ταχύτητας επιβατικά πλοία, ε, τρένα. Δεν αρκεί λοιπόν αυτή η γραμμή. Και επίσης χρειάζεται ουσιαστική βέλτιωση της διαλειτουργικότητας του διαδρόμου για να ενισχύεται η μεταβίβαση, η μεταφορά στη σύγχρονη τεχνολογία, μήκος σειρμού, συστήματα σημάτων, φορτίο άξονα. Για δε την Ισπανία χρειάζεται μετατροπή των ε, ιστορικών γραμμών που χρησιμοποιούνται για, τον, ε, ε, για τα φορτία κυρίως από τον Ιβυρικό στον ευρωπαϊκό, στο ευρωπαϊκό πρότυπο. Μικρό μόνο ποσοστό των μεταφορών από την Ισπανία μέχρι την Ιταλία γίνονται σιδηροδρομικό, στο μεγαλύτερο κομμάτι είναι ε, ναυσιπλοϊκό, αλλά και οδικές μεταφορές φορτίων. Δαπανηρό, αλλά και μη βιώσιμο σύστημα. Επίσης, Πρόεδρε, οι νέοι διαδρομή TNT πρέπει να είναι πολυλειτουργική. Και έτσι έχουμε το κομμάτι του τελευταίου μιλίου ή χιλιόμετρου και τη διασύνδεση με βιομηχανικές περιοχές και δυνατότητες μεταφόρτωσης που χρειάζεται ιδιαίτερη υποστήριξη. Έχουμε 30 μίζωνες λιμένες που πρέπει να συνδεθούν με τη χώρα. Ύστερα από μια σύντομη επισκόπηση, στρέψτε μου τώρα να φερθώ στις προτεραιότητες που θέλω εγώ να ορίσω για τον Μεσογειακό Διάδρομο. Πέντε, καταρχάς τα σημεία κλειδί να, η διασύνδεσης να ολοκληρωθούν όπου λείπουν. Ε, το τωρινό Λιόνε παραδείγματι είναι ο άξονας από τον οποίο θα εξαρτηθεί η λειτουργία του άξονα, γιατί δεν θα υπάρχει διαφορετικά διασύνδεση μεταξύ ανατολικού και δυτικού τμήματος του άξονα νοτίως των Άλπαιων. Αυτό είναι το σημείο κλειδί. Ε, δεύτερον, το Μομπελιέ Περπινιό χρειάζεται να αναπτυχθεί για να εξασφαλίσει το πλήρες δυναμικό του άξονα, όπως είπα νωρίτερα, αλλά αυτό ισχύει και για το ανατολικό κομμάτι, διασυνοριακό, ε, δηλαδή συνοριακές μεταφορές, και ιδιαίτερα καθώς πρόκειται για χώρες συνοχής προς Ανατολάς θα έχει σημαντικό κομμάτι για τη συνοχή αυτό. Τρίτον, διαλειτουργικότητα. Διαφορές ε, ε, προτύπων ανέφερα ήδη νωρίτερα, ε, αλλά υπάρχουν και πολλά άλλα προβλήματα που πρέπει να καλυφθούν. Τέταρτος στόχος, διασύνδεση των κυρίων θαλασσίων λιμένων με την ενδοχώρα και έτσι πρέπει να ολοκληρωθεί η διασύνδεση με τις οδικές και τις ιδιοδρομικές μεταφορές και τους λιμένες. Το επόμενο θέμα το περνάω γιατί καλύφθηκε, αλλά το τελευταίο, τελευταία προτεραιότητα ανάπτυξη δηλαδή των αστικών κόμβων έχει πολύ μεγάλη σημασία και αυτό όχι μόνο για τις επιβατικές μεταφορές αλλά και για τα φορτία με την ίδια σημασία. Είναι αξιόλογο το γεγονός ότι δεν είναι επαρκώς ε, ανεπτυγμένη η αστική κόμβη μέχρι σήμερα. Κλείνοντα, πρόεδρε, θέλω να πω ότι χρειάζεται να αλλάξουμε νοοτροπία στην Ευρώπη. Πρέπει να αλλάξουμε από την εθνική προοπτική στην προοπτική την ευρωπαϊκή. Η ευρωπαϊκή προοπτική είναι το κύριο στοιχείο ε, με το οποίο μπορεί να προχωρήσει αυτός ο μεσογειακός άξονας και τα υπόλοιπα είναι ε, αυτά, εξαρτώνται από αυτήν. Ευχαριστώ πολύ, λέει ο Πρόεδρος. Ερωτήσεις. Αγιάλα Σέντερ. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Μπριγχόρστ για μια παρουσίαση Πρέπει να ξαναξεκινήσετε γιατί προσπάθησα να κλέψω τα ακουστικά του Προέδρου, λέει ο κύριος Μπριγχόρστ. Θα ήθελα λοιπόν να σας ευχαριστήσω κύριε Μπρίγχορστ για την παρουσίασή σας αυτή της πρώτης έκθεσης με στοιχεία ουσιαστικά μελέτης, γνώσης για τη μοναδικότητα και τα προβλήματα της περιοχής, όπως επίσης και για το ότι αναγνωρίζετε ότι είναι ανάγκη να λύσουμε κάποιες, κάποια από τα σημεία συμφόρησης. Σας ευχαριστώ που ήσασταν τόσο ειλικρινείς. Και είπατε στην αρχή πως το ευρωπαϊκό οικοδόμημα είναι κάτι που εναντιώνεται στη φύση και καλό είναι να περάσουμε την αδράνεια των κρατών μελών που προστατεύουν σαν τρελά τα εδάφη τους και τις επιχειρήσεις τους και τις δικές τους υπηρεσίες. Είμαστε στην περιφέρεια και όσοι είμαστε εκεί αντιμετωπίζουμε διπλά και τριπλά προβλήματα για να καταφέρουμε να φτάσουμε στο κέντρο της Ευρώπης. δεν φαίνεται από εδώ καλά, αλλά στην πρόταση που κάνετε του χάρτη εδώ, εγώ πάντα έχω πρόβλημα με τους χάρτες και γι' αυτό ε, αντιμετωπίζω πάντα πρόβλημα και εδώ και αλλού. Πάντως σίγουρα φτάω γιατί βλέπω κάποιες γραμμές πιο σκούρες, άλλες πιο ανοιχτόχρωμες αλλά νομίζω πως αυτή η διαδρομή της Μεσογείου που φεύγει από το Αρχεσίρας και φτάνει σε δύο τμήματα στο βορρά, περνώντας από το κέντρο της ε, Ισπανίας, είναι ένα τμήμα που φτάνει στη Σεβίλη, που είναι ε, λιμάνι σε ποτάμι, και μετά θα πρέπει να ενώσει την Ανδαλουσία με την Αλμερία. Αυτό δεν το βλέπω στο χάρτη γιατί βλέπω την Αλμερία, τη Μούρσια που είναι ε, και την Καρταχένα που είναι πιο βόρεια, αλλά κάπου θα έπρεπε να υπάρχει και μια γραμμή που να συνδέει με την ε, αριστερή πλευρά την Ανδαλουσία. Το λέω, είναι τόσο ανοιχτό χρώμα που δεν φαίνεται. Γιατί η διαφορά είναι το πρώτο που θα κοιτάξουν στην Ανδαλουσία και καλό είναι να διατηρηθεί αυτό. Είναι ένα από τα ουσιαστικά σημεία του διαδρόμου ενώνει το λιμάνι του Αλχεσίρας με το λιμάνι της Μαδρίτης που βέβαια είναι ένα ξηρό λιμάνι αλλά εκεί πάνε περισσότερα ψάρια που και είναι η μεγαλύτερη αγορά αλλιεύματος και συνεχίζει μετά παράλληλα με τη Μεσόγειο. Σας ρωτώ επίσης το εξή. Υπάρχει μία παραδοχή στην Ισπανία που λέει το εξής. Είμαστε μια παράδοξη χώρα, είμαστε μια χώρα η οποία ήταν σε απομόνωση, όπως και οι χώρες της Βαλτικής. Ίσως λοιπόν καλό θα ήταν να χρησιμοποιήσουμε τις δυνατότητες που δίνουν τα απομονωμένα δίκτυα. Γιατί πολλές φορές με τις εμπορευματικές συνδέσεις επειδή ακολουθήσαμε το μοντέλο της υψηλής ταχύτητας με τρένα που τρέχουμε πάνω από 300 χιλιόμετρα, έχουμε απελευθερώσει, γιατί αυτό το έχουμε διαθέσει στους επιβάτης, την παραδοσιακή ισπανική γραμμή ε, στα επορεύματα. Και βέβαια όταν φτάσουν στα σύνορα υπάρχει πρόβλημα. Ξέρετε πως τα δύο συνοριακά περάσματα ε, χρειαζόταν αλλαγή αξονίου αυτό το έκανε η Τρανφέσα, την αγόρασε η Deutsche Bank και αυτή τη στιγμή το πρόβλημα που έχουμε στα σύνορα είναι πώς θα καταφέρουμε να γίνεται ακριβώς αυτή η αλλαγή. Επίσης, η λύση, η τρίτη, που είναι να κάνουμε αυτή την αλλαγή από τις παλιές ε, γραμμές στις τροχές που έχουν την, ε, το ευρωπαϊκό πλάτος ανοίγματο είναι μια δυνατότητα, αλλά στις περιφερειές που, που εφαρμόζεται αυτό, παρόλο που ήταν μια καλή λύση για να λύσουμε το πρόβλημα της Καταλωνίας προς το Βορρά και τη Γαλλία, ε, δεν ε, περνάει σαν κάτι θετικό. Δηλαδή αυτή η τρίτη λύση ε, με την τρίτη γραμμή που προσθέτουμε δίπλα στις άλλες δύο θεωρείται κάπως ε, μειονεκτική. Υπάρχει τρόπος αυτό να το λύσουμε. Και θα κλείσω αυτό, μην ανησυχείτε πρόεδρε, για τη διαλειτουργικότητα και την αλλαγή και τα πολυμέσα. Ε, υπάρχει πρόβλημα και με τα τούνελ στη Νότια Ευρώπη γιατί εκεί υπάρχει μια απλή λύση, επειδή το ύψος δεν είναι παρκές, να έχουμε πιο χαμηλά βαγόνια. Αλλά δυστυχώς αυτά δεν τα βρίσκουν οι εταιρείε. Δεν έχουν αρκετά τέτοια οι φορείς, οπότε ίσως θα έπρεπε το θέμα αυτό να το συμπεριλάβουμε ως λύση για να εξασφαλίσουμε τη διαλειτουργικότητα. Ο Ντομινίκ Ρικέ, επόμενος ομιλητής. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ τον κύριο Μπρίνχορστ για την παρουσίαση που έκανε. Έχω δύο ερωτήσεις για δύο τμήματα που με ενδιαφέρουν πιο πολύ. Είπατε πρώτα απ' όλα πως υπάρχει ενδιαφέρον αλλά και δυσκολία για το Περπινιάν Μομπελιέ. Ξέρω πως εκεί υπάρχουν δύο ενδεχόμενες διαδρομές, μία η οποία ακολουθεί την ακτογραμμή αλλά και έχουμε περιβαλλοντικά προβλήματα και έχει μεγάλες πληθυσμαστικέ ομάδες και άλλοι που θα περάσει από τα βουνά Κορμπιέρα, από την οροσύρα εκεί, αλλά βέβαια το κόστο είναι υπέρογκο. Υπάρχει εκεί κάποια επιλογή που να έχει γίνει ή βρίσκεται πάντα σε κρεμότητα το θέμα και δεύτερον. Για, για το Λιόν Τορίνο πάντα μιλάμε για το τούνελ της Τουντέλα, αλλά εγώ δεν το σκέφτομαι αυτό, μιλάω για την προσβασιμότητα γενικότερα. Υπάρχουν δύο θέματα που έχουν προκύψει και είναι σε κρεμότητα αυτή τη στιγμή. Το αν θα υπάρξει παρακαμπτήριος δακτύλιος για το νότιο-ανατολικό κομμάτι της Λιών επρόκειτο να χτιστεί με κόστος 600 εκατομμύρια ευρώ αλλά τελικά χρησιμοποιείται μία γραμμή η οποία δεν είναι αρκετά καλή. και όπου χρειάζεται γύρω στα 20 δις εργασίες ε, για τα 40 δις στα, οποία αναφέρθηκα προηγουμένως γίνεται αυτή, αυτή τη στιγμή κάποια διαιτησία έτσι ώστε να γνωρίσουμε ποιο θα είναι το χρονοδιάγραμμα της χρηματοδότησης κτλ για τα δύο αυτά τμήματα τα οποία είναι πάρα πολύ σημαντικά για να συνδέσουν την Ισπανία και την Ιταλία και να απελευθερώσουμε και τον, ε, νότιο, και τον, βορρά, με και τον άξονα βορρά-νότου. Ο κύριος Σαλίνη. Grazie. La, diciamo, la premessa che ha, che ha posto è... Πάρα πολύ σαφή τα όσα μας είπατε όσον αφορά και αυτή την πλαισίωση αυτού του είδους τη, σημασία αυτού του διαδρόμου. Αλλά έχουμε κάποια στατιστικά στοιχεία. Πολύ είναι σχετικά, διότι ο ρόλος αυτού του διαδρόμου όσον αφορά την οικονομία μας είναι κάτι το οποίο έχει συνέπειες που ε, ε, ε, οι συνέπειες είναι, είναι ανάλογα με τον κάθε τομέα που θέλει να εξετάσει και όπως μας είπατε έχουμε κάποιους κόμβους. Έχουμε επίσης κάποια έλλειψη διασυνδέσεων με τον σιδηρόδρομο. Ε, ε είπατε αλλού έχουμε διασυνδέσεις με λιμάνια και όχι με αεροδρόμια, Φερρυπίν. Άρα, τι θα γίνει με την κυκλοφορία των επιβατών. Είπατε για το 20% σε Κροατία και Σλοβενία. Επομένως, αυτός ο διάδρομος ε, χαρακτηρίζεται από την ανισότητα για τα προβλήματα στη διασυνδεσιμότητα και εμάς ε, η διασύνδεση του Τωρίνου με την Λιόν είναι πάρα πολύ σημαντικό οικονομικά. Μιλάμε για το 30% των εισαγωγών μας πέραν από εκεί. 64 δις ευρώ αξίζουν αυτά τα εμπορεύματα και μιλάμε για 85 ε, δισεκατομμύρια εξαγωγές που στέλνουμε και επομένως και εδώ έχουμε για αυτή τη διαδρομή ε, πολλά αντιεπιχείρηματα, πολλές αντιρρήσεις και ενστάσεις. Ακριβώς όπως ανέφερε εν μέρει και ο κ. Θέλω τώρα άλλα τρία στοιχεία να προσθέσω. Ίσως είναι σημαντικά ο χαρακτήρα. Πρώτα πρώτα για την διασύνδεση ε, και τη σχέση του διαδρόμου με το πρόγραμμα Juncker. Γιατί είπαμε ότι πόσο σημαντικό είναι να έχουμε κάποιες επενδύσεις στους διαδρόμους που να καλύψουν και αυτόν τον διάδρομο. Οπότε το ερώτημα από αυτό είναι το εξή. Στο πλάνο, στο σχέδιο Juncker θα πρέπει να δούμε πότε και πόσο θα μπορέσει να υποστηρίξει τις επενδύσεις πρέπει να γίνουν για τα τρένα. Ε, η απάντηση φυσικά και είναι δύσκολη, αλλά ο διάδρομος για τη Μεσόγειο σε σχέση με τη, τη δέσμη των τηλεδρομικών μέτρων ε, αναδεί πολλά ερωτήματα. Τώρα κάτι άλλο. Ε, ξέρουμε ότι έχει προγραμματιστεί μία διεύρυνση της διόργας του ΣΟΕΣ. Αυτό άμεσα θα έχει συνέπειες στις ισορροπίες που θα περτανεύουν στη Μεσόγειο. Γιατί επομένω <clears throat> μπαίνουμε στη λογική αυτού του διαδρόμου χωρί να λάβουμε υπόψη αυτό που θα γίνει στο Σουέζ. Κάτι άλλο τώρα. Η Μεσόγειος είναι το σημείο στο οποίο περνάνε οι μεταναστευτικές ροές. Ε, τώρα επομένως θα πρέπει αυτή την προβληματική ε, να την λάβουμε υπόψη όσον αφορά τις επενδύσεις για τον ε, διάδρομο. Γιατί πρόκειται για μια άλλη ροή. Ε, οπότε θα πρέπει να δούμε πώς αυτό θα επηρεάσει τις χώρες που βρέχονται την Μεσόγειο. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Κύριε Στονιστή. Μια πολύ μεγάλη τρύπα βλέπουμε στο χάρτη. Δυτικά Βαλκάνια. και μία από τις κύριες ε, πτυχές προσέγγισης Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, στην προσέγγιση της μετακράτη αυτά είναι ακριβώς η συνδεσιμότητα. Ο Επίτροπος Χάν και η κυρία Μπούρτς και οπότε έχει γίνει συζήτηση για τις έξι αυτές χώρες Νοτικών Βαλκανίων εν γέννη υπογραμμίζεται ότι Εκείνοι οι κύριοι δρόμοι, οι κύριες διαδρομές που φτάνουν στις χώρες αυτές πρέπει να διασυνδεθούν μεταξύ τους μέσω των ευρωπαϊκών δικτύων. Στην πρώτη αναθεώρηση θα δούμε τι μπορεί να έχει γίνει εντωμεταξύ και ρωτώ τον συντονιστή τι σχόλιο έχει γενικά για την πολιτική αυτή, για τη διασύνδεση των Βαλκανίων των Δυτικών Βαλκανίων. Τι γίνεται για την περιοχή αυτή που γεωγραφικά ανήκει στην, Ευρώπη, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και επίσης, πότε νομίζω ότι θα γίνει αυτή η αναθεώρηση του δικτύου Τέντη. Ο πρόεδρος, ευχαριστώ κύριε Σφαντάν Κάμπ. Ε, ευχαριστώ πολύ πρόεδρε. Νομίζω ότι διάλεξε το διάδρομο με, με τις καλύτερες κοινοτολογικές συνθήκες και με τις ωραιότερες παραλίες ο κύριος Στενιστής. Έχω λοιπόν τις εξής ερωτήσεις. Έχουμε μία στροφή μοντέλου. Μιλούμε για διαλειτουργικότητα και σύνλειτουργικότητα. Αλλά δεν φαίνεται να μπορούμε να ξεφύγουμε από τι οδικέ μεταφορέ. Πώ μπορούμε να πιέσουμε γι' αυτό, έχετε κάποιο όραμα. Είναι πολύ μεγάλα το μερίδιο των οδικών μεταφορών σε αυτό το διάδρομο. Η σύραγγα. Λιόν Τουρίνου. Ρήνου. Είναι τιτάνιο έργο. Πώς έχει προχωρήσει. <coughs> το θέμα δεν είναι μόνο το χρήμα, είναι οι άδειες, ε, οι περιβαλλοντικές ζημιές, όλα αυτά είναι υπό έλεγχο ώστε να τηρηθούν και τα χρονοδιαγράμματα. Τρίτον, επενδύσεις από τους Κινέζους. Άλλοι τις θεωρούν ε, ευκαιρία, άλλη απειλή. Εσείς τι λέτε για τους Κινέζους και τα κεφαλαία τους. Και εάν μου επιτρέπετε να είμαι και λίγο θρασής, η συνεργασία μεταξύ γαλλικής και ισπανικής κυβέρνησης στο διαδρομό σας. Δεν έχετε περιθώριο να τη βελτιώσετε. Ο πρόεδρος έχει σε μια θρασία ερώτηση, θα λάβετε και θρασία απάντηση φαντάζομαι. Η Καριμάντελή όμως. Έχει πρώτο το λόγο. Αγαπητή συνάδελφοι, κύριε Μπρίνκχορστ, σας ευχαριστώ πολύ για αυτή την παρουσίαση. Νομίζω ότι όλοι χαμογελάσατε όταν ακούσατε Λιόν Τωρίνο. Επανέρχομαι σε αυτό, αν σας κατάλαβα καλά. Και θέλω να μου το επιβεβαιώσετε. Αυτό το τούνελ των 57 χιλιόμετρων μπορείτε να επιβεβαιώσετε πως ολόκληρο θα κοστίσει 26 δις. Alors, quand on Mm. Όταν... Αυτό θα μου πείτε. Θα μου πείτε, δεν ζητάμε από την Ευρώπη, από την Ευρώπη να χρηματοδοτήσει ολόκληρο το έργο, ένα τμήμα. Και όταν βλέπω πως η Ευρωπαϊκή Ένωση θα συνεισφέρει το 40% αυτού του προπολογισμού, μιλάμε για 12 δις. Για ένα τούνελ, μία σύραγγα. Ρωτώ λοιπόν. Μια και μειώνουμε αυτή τη στιγμή το μηχανισμό ολόκληρο ε, της διασύνδεσης της Ευρώπης, τι θα κάνετε. Και επίσης, αν το 40% το βάλει η Ευρώπη, είστε βέβαιοι ότι η Γαλλία και η Ιταλία που αυτή τη στιγμή έχουν δυσκολίες σε οικονομικό επίπεδο, σας έχουν επιβεβαιώσει πώς θα αναλάβουν την οικονομική βιωσιμότητα του 60% αυτού του προπολογισμού. Δεύτερη ερώτηση. Μου είπατε πως είστε υπέρ της πολυμεσοτικότητας. Μα ποιος είναι εναντίον. Όλοι θέλουμε αυτή τη στιγμή τα φορτηγά να τα φορτώνουμε ε, σε βαγόνια. Όποιος διαφανεί να σηκώσει το χέρι του. Αλλά το έργο θα πρέπει να κλείσει. Πότε θα τελειώσει αυτό το έργο. Έχετε κάποια προθεσμία. Το 2030 θα έχει χτιστεί. Θα περιμένουμε δηλαδή να λύσουμε το θέμα των κόμβων και της ρήπανσης το 2030 από σήμερα. Το θέμα της ρήπανσης και του κλίματος έχει να κάνει με τις μέλουσες γενιές. Οπότε ρωτώ, μήπως δεν υπάρχουν κάποια εναλλεκτικά σχέδια Μήπως έχετε μελετήσει κάποιες άλλες αναλεκτικές λύσεις εκτός από αυτό το περίφημο Λιόν Τωρίνο. Επίσης, η Ιταλία και η Γαλλία θεωρούν σήμερα πως θα μπορέσουν να το χρηματοδοτήσουν μέσω του σχεδίου Juncker. Θέλω και εδώ συγκεκριμένη απόφαση. Και τέλος, όποιος διάδρομος και να είναι, υπάρχει ένας κανόνας είναι βαρχίδα των κανόνων που είναι ο εξή. Οι πολίτες ερωτήθηκαν. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Θα αναφερθώ και εγώ στο σχέδιο και αφενός μεν λόγω της εμπειρίας που έχω από άλλα σχέδια και έργα και ακούσαμε ότι οι προτεραιότητες είναι το σουιοδέστερο Ακούω ότι έχει οικονομικά προβλήματα η γαλλική κυβέρνηση και άρα η γραμμή Μπορτό Μπιλμπάο καθυστερεί. δεν θα κατασκευαστεί τα επόμενα χρόνια γιατί δεν έχει τα σχετικά κονδύλια να διαθέσει η Γαλλία. Όταν το γαλλικό δε ελεγκτικό συνέδριο είπε ότι το Λιόν Τωρίνο δεν θα κοστίσει 12 αλλά 26 δις, ο Μόντι και ο Λόντ ήρθαν και είπαν «Α, τι, δεν τίποτα, 14 πλέον δισεκατομμύρια θα τα δώσει η, η Ευρωπαϊκή Ένωση». αυτό δεν υπάρχει καν το χρήμα, δεν υπάρχει θέμα δηλαδή να διατεθεί. Άρα δεν θα έπρεπε να υπάρχουν προτεραιότητε και δεν υπάρχουν και πιο σημαντικά σημεία διασύνδεση. Στον Πορτό για μένα είναι πολύ πιο σημαντικό γιατί η Ισπανία έχει κάνει τεράστια βήματα πρόοδου σε σχέση με την υλοποίηση, ε, την εισαγωγή των ε, τρένων υψηλή ταχύτητα. Μεγάλο επιτεύγμα και για την Ισπανία αλλά και για την Ευρώπη μεγάλο κέρδο και γι' αυτό είναι σημαντικό, πολύ πιο σημαντικό για μένα να δοθεί προτεραιότητα σε αυτό. Σχόλια χωρίς μικρόφωνο από την κυρία Γιάλα Σέντερ. Ήμασταν στο Βιλμπάο. Και εκεί μας είπανε, ναι, ναι, το ξέρω, αλλά είπανε ότι το τρίγωνο του Ατλαντικού είναι στην συνήθη γραμμή, την παραδοσιακή γραμμή και πρέπει να βελτιωθεί για να έρθει διασύνδεση. Όλα αυτά μας είπανε. Ε, ρωτώ λοιπόν, αυτή θα είναι η μόνη διασύνδεση νοτίως των Αλπέων Μα προφανώς υπάρχουν και άλλες δυνατότητες, υπάρχουν και οι ακτογραμμές και υπάρχουν και άλλες γραμμέ ε, δεν μπορεί να ισχυριστεί κανεί ότι δεν είναι συνδεδεμένο το, το ρήνο με τη Λιόν αυτή τη στιγμή, γιατί η γραμμή υπάρχει, απλώς χρειάζεται εξυγίανση και αν πρόκειται να κοστίσει άλλα 16 δισεκατομμύρια το έργο τη σύραγγα, α κάνουμε την ανάλυση ποιο είναι το πιο οικονομικά συμφέρον έργο και σε αυτό να δώσουμε την έμφαση. Άλλωστε θα πάει και πιο γρήγορα, θα είναι και πιο αποτελεσματικό αφού υφίσταται ήδη η γραμμή. Εάν χρειαστεί λοιπόν 30 χρόνια αυτό το... αυτή η σύραγγα, μακάρι να είμαστε όλοι, ε, να γίνουμε όλοι υπεραιωνόβιοι και να ζήσουμε να το δούμε, αλλά δεν φαίνεται. Αυτό είναι που δεν υπάρχει στην Ευρώπη. Διασύνδεση μεταξύ Βερολίνου, μάλλον Αμβούργου, ε, Βερολίνου, Μπρέσλαου, Κράκοβιτς, μια γραμμή στην οποία λείπουν από το Κότπους μέχρι τα σύνορα της Πολωνίας 50 χιλιόμετρα, μια γραμμή σιδηροδρομική για την οποία θα χρειάζονταν 100 μόνο εκατομμύρια για να καλυφθούν τα τελευταία αυτά 50 χιλιόμετρα της σιδηροδρομικής γραμμής. Και για να δώσω και ένα γερμανικό παράδειγμα, Μπορεί να δώσουμε 10 δισεκατομμύρια για να κερδίσουμε 30 λεπτά μόλις χρόνο σε Στουτχάρδη. Ε, λοιπόν, ε, γιατί να χρειαστεί να χάσουμε τόσο χρόνο για τη σύραγγα του Τωρίνου, γιατί να, μιλήσουμε, να μιλήσουμε το πρόβλημα υφιστάμενα ή με άλλα έργα τα οποία είναι πιο γρήγορα και πιο οικονομικά και γιατί να μην γίνει η έρευνα με βάση τα όσα είπε το ελεγκτικό συνέδριο ότι δεν θα κοστίσει 12 αλλά 26 δις και να επαληθευθούν οι εναλλακτικές. Γιατί να εμένουμε να κάνουμε αυτό το έργο το τόσο, ε, το τόσο, το, τόσο δαπανηρό και το τόσο, τόσο χρονοδοβόρο. Έχετε πολλές ερωτήσεις λοιπόν, να απαντήσετε κύριε Μπρίνκχορστ. Πάντοτε είναι ευχαριστώ για μένα να έρχομαι εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, γιατί όπως ξέρετε διατέλεσα Ευρωβουλευτής και έχω ακόμα το μπάτζι το οποίο περήφανα το κρατάω για την 94-99. Ε, Τώρα βέβαια είναι πιο δύσκολο κανείς να εκλεγεί, είναι σαν να μπει μάλλον στο κοινοβουλίο, ε, σε έχει γίνει φρούριο. Τέλος πάντων, εγώ σαν συντονιστής είναι το να δούμε κατά πόσον εσείς μπορείτε να βελτιώσετε την ευκολία να μπει κανένα στο κτίριο. Ε, εντάξει, εγώ έκανα 25 λεπτά να, για να έρθω εδώ και να μπω, να φτάσω στην αίθουσα. Αλλά τι, θα, τι να κάνει ο Κοσμάκης, πώς θα μπει, τι γίνεται με την διαφάνεια, τέλος πάντων. Πρόεδρε, πάντοτε η ευθύτητά σας με ενθουσιάζει και τώρα για να απαντήσω πρώτα-πρώτα στην κυρία Αγιάλα Σέντερ. Κοιτάξτε, έχω εδώ πέρα αυτό το φύλλο, αυτό το χάρτη. Ε, βέβαια είναι αρκετά γενική άποψη, αλλά δεν, δεν, δεν, δεν θυμάμαι τι γίνεται με την Ανταλουσία. Φυσικά είναι πάρα πολύ σημαντική για την Ισπανία και φυσικά θα υπάρξει εκεί πέρα ε, κάποια σύνδεση με τον ε, διάδρομο της ε, Μεσογείου. Και θα σας πω σε λίγο για το στατικό χαρακτήρα του διαδρόμου. Όταν μιλήσω στην κυρία από τη Γαλλία, εδώ εξ αριστερών. Οπότε, ε, αν υπάρχουν κάποιες επιφυλάξεις, κάποιες αμφιβολίες για το πρόγραμμα εργασιών, θα σας ενημερώσω εγγράφος. Φυσικά και πρέπει, αν έχετε τέλο πάντων τώρα αμφιβολίες, θα, θα σας τα πω γιατί είναι σημαντικό τώρα. Το θέμα της λύσης για την πύλη. Για την Ισπανία η οποία έχει κάνει πολύ περισσότερα από όσα για το μέγεθος της, ε, της τροχιάς ε, έχετε κάνει αυτά που πρέπει για να περάσει το τρένο και νοτίως των Πυρηναίων και βεβαίως ε, θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό ε, αυτό γιατί ε, κάποτε λέγαμε ότι θα πρέπει να είστε κλεισμένοι με τα Πυρηναία αλλά αυτό δεν είναι ευρωπαϊκή λύση άρα θα πρέπει η, η απόσταση αυτή των γραμμών να βελτιωθεί, να προσαρμοστείτε. Άρα αυτό Επίση, θα, να δούμε τι θα γίνει με τις σύραγγε, κατά πόσον έχουμε το θέμα του ύψου τη σύραγγα. αν θα πρέπει να μειωθεί. Δεν είμαι μηχανολόγο, αλλά θα πρέπει να καταλήγουμε στο ότι μάλλον δεν χρειάζεται, γιατί έχουμε και τα τρένα που μεταφέρουν containers. Το είπε και ο πρόεδρος σωστά, γιατί νοτίως των Άλπιων υπάρχει ο διάδρομος και έχουμε κύριε Κράμε 200 σύραγγες μεταξύ της Νίκαιας και της ε, Γένοβας. 200, 200 τούνελ. Οπότε να προσαρμόσουμε 200 τούνελ για να μπορούν να χωρέσουν αυτά τα κοντέινερ είναι τεράστιο, αστρονομικό. Οπότε, τι να σας πω, δεν ξέρω πώς θα κόστιζε η προσαρμογή των ισπανικών σειράγκων. Θα το μελετήσω και θα σας πω, αν γίνεται. Βεβαίω και πρέπει να υπάρξει διάλογο μεταξύ μα. Αλλιώ η απάντησή μου δεν είναι απάντηση. Κύριε Πίκη, θα ήθελα να σα τα πω στα γαλλικά, αλλά δεν θα καταλάβαιναν οι άλλοι τόσο καλά. Επομένω, θα συνεχίσω να τα λέω στα αγγλικά. Επιλέξτε, επιλέξτε ότι εγώ τη γλώσσα δεν μπορώ να μιλήσω, λέει ο Πρόεδρο. Τέλο πάντων, στο παρελθόν είχα ζωήσει πολύ του διερμηνεί μίλαγα στο Συμβούλιο των Υπουργών σε ε, γλώσσα άλλη από την Ολλανδική. Και μου λέγανε κύριε Υπουργέ καλύτερα μιλήσετε τη γλώσσα σας. Οπότε έτσι και εγώ προσαρμόστηκα. Τέλος πάντων για την σύνδεση Περπινιάν Μονπελιέ. Κύριε Ρικέ, έχω να σας απαντήσω το εξή. Εξαρτάται από την γαλλική κυβέρνηση να προσαρμόσει το πρόγραμμα εργασιών. Εμείς έχουμε καταρτήσει ένα πρόγραμμα αυτό που ισχύει, το ενέκριναν όλα τα κρατημέλη, όλες οι μη κυβερνητικέ οργανώσεις και όλες οι περιφέρειες και οι άλλοι εμπλεκόμενοι. Δεν μπορώ να σας πω για εναλλακτική λύση. Και αυτό που είπαμε και ισχύει για την Ισπανία είναι ότι μετά το Λιόν του Τωρίνο θα φροντίσουμε να γίνει και η προσαρμογή ε, της διαδρομής Μομπελιέ ε, Περπινιάν. Οπότε έτσι θα πρέπει να υπάρχει πρόσβαση στην υπόλοιπη Ευρώπη. Είπαμε ποια είναι η εθνική διάσταση της υπόθεσης. Αλλά θα πρέπει επίσης να γίνει κατανοητό το ότι έχει στρατηγική διάσταση ο διάδρομος αυτός. Και επίσης συνδέεται με τους άλλους οκτώ διαδρόμους και αν δεν συνδέεται δεν θα λειτουργήσει υπόθεση. Δεν είναι θέμα μόνο επομένως ε, το κόμμα μου Πελία Περπενιά. Οπότε παρακαλώ ε, επευθυνθείτε στη γαλλική κυβέρνηση. Αυτοί να επιταχύνουν το ρυθμό τους. Σύντομα πιστεύω ότι θα υπάρξει διάλογος ε, Γαλλίας-Ισπανίας όπως έγινε τόσα χρόνια τώρα, 8 χρόνια τώρα μεταξύ Γαλλίας και Ιταλίας. Άλλα 5 λεπτάκια. Και μετά πρέπει να τελειώσω. Πρέπει να είμαι τότε πάρα πολύ σύντομος γιατί μόνο σε εσά να απαντήσω μου πήρε μισή ώρα. Μόνο μισό ο πρόεδρος. Ε, ο πρόεδρος προηγείται. Τέλο να θα είμαι πάρα πολύ σύντομο. Ξανά και ο Μπρίγχος. Τώρα, όσον αφορά την παρακαμπτήρια για τη Λιόν και την σχέση Λιόν Τωρίνο. Σε 12 χρόνια, όχι σε 30, σε 12 χρόνια θα έχει ολοκληρωθεί αυτή η σχετική σύραγγα. Ελπίζω να ζήσω για να το δω. Και κύριε Ανταλή, τότε θα είναι απλώς με σύλληβε αυτό. Οπότε, το θέμα είναι το ότι στο μεταξύ θα πρέπει να συνεργάζεται και η γαλλική κυβέρνηση. Αλλά αυτό είναι κάτι το οποίο επισημαίνεται στο πρόγραμμα εργασία. Δεν μπορώ να το σχολιάσω τώρα. Κύριε Σαλίνη, βεβαίως είναι πολύ σημαντικό και για την Ιταλία το έργο. Και ξέρετε είχαμε από δεξιά και από αριστερά αντιρρήσεις επί πέντε διαδοχικές κυβερνήσεις για τις Άλπες. Είπατε κάτι για το πρόγραμμα Γιούνκερ και εσείς όμως κύριε Πρόεδρε. Όχι, δεν υπάρχει συγκεκριμένη διασύνδεση. Το σχέδιο Γιούνκερ χρηματοδοτείται εν μέρη από χρηματοδοτήσει εν μέρη τι μεταφορέ, Εν μέρη. Το είπαν και στην Και βέβαια θα καλυφθεί, θα ωφεληθεί από τον διάδρομο το σχέδιο Γιούνκερ. γιατί βέβαια θα τονωθεί η οικονομία, θα υπάρχει καλύτερη επιμελητία και φυσικά ξανοίγονται προοπτικές επενδύσεων. Τώρα για, το, τη διόρυγα του Σουέζ που είπατε κύριε Σαλίνη, αλλά και ο κύριος Φαντεκάμπ αναφέρθηκε, ιδίω η Μεσόγειος θα ωφεληθεί. Όπως λέω εγώ τα πράγματα προσωπικά δεν είναι θέση της Κομισιόν η εμπλοκή δηλαδή, και των Κινέζων και αυτά δεν υπάρχουν στην έκθεση. Υπάρχει εδώ μια στρατηγική διάσταση. Να πάει κανείς από Κίνα στην Ευρώπη. Φτάσει στη Μεσόγειο. Και κανείς έρθει γύρω-γύρω από την Ισπανία αυτές τις τέσσερις μέρες. Άρα θα πρέπει να βελτιωθούν οι λιμένες. Ευτυχώς αυτό τώρα δεν είναι επίκαιρο, δεν, είναι, δεν χρειάζεται να γίνει άμεσα. Αλλά σε συνεργασία με τους αδελφούς που ασχολούνται με τους λιμένες θα δούμε το πώς θα συνοηθούμε με τα πέντε λιμάνια. Ραβένα, Βενετία, Τωρίνο, Ριέκα και γιατί θα συνεργαστούν αυτοί οι λιμένες όσον αφορά την προσβασιμότητα. Θα είναι βέβαια και εναλλακτική του Ρότερνταμ αυτή η, η ρύθμιση και να με συμπαθάει ο πρώην πρόεδρος της Ολλανδίας γιατί προς το παρόν είναι μηδενική συνεργασία. το λέω αυτό και στον συνάδελφο από την Κροατία. Γι' αυτό και θέλουμε το Κοινοβούλιο να βοηθήσει και να αναδείξετε αυτήν την στατική διάσταση των εξαγών της Κίνας και των επενδύσεων των Κινέζων. Είναι στρατηγικά αυτά τα λιμάνια, ιδίως όσον αφορά την Κίνα. Είχα πεντάλει το πρόεδρο, αλλά θέλω να πω δύο λόγια στην κυρία Κάρμανταλή και σε εσά. Αλλά πρώτα πρώτα. Εσείς από την Κροατία είστε το πιο πρόσφατο μέλος, αλλά καλύπτεστε από τον διάδρομο. Δεν μπορώ τώρα να το αναλύσω, αλλά δούμε, θα, θα πάω στη Ριέκα, πήγα στο Ζάγκρεπ, οπότε η σύνδεση είναι άριστη Ουγγαρίας, Σλοβενίας, Κροατίας και είναι χώρε συνοχής, συνάντησα τους υπουργού και των τριών χωρών. Δεν μπορούμε από τώρα να, να, πούμε τι θα γίνει με Σερβία, Μαυροβούνια κλπ. Αλλά από ό,τι θυμάμαι η αυτοτρία των Αψβούργων είχε τη Ριέκα ως βασικό λιμάνι. Άρα αυτό σας δείχνει την σημασία και την ιστορία του λιμένου. Τώρα, για να δούμε, κύριο Φαντεκάμπ τον εκάλυψα, αλλά θα πρέπει να τα πούμε οι δυο μας όσον αφορά το συνδυασμό των μεταφορικών μέσων κλπ. Αλλά πρώτα δεν με αφήνει να το αναλύσω. Κυρία Καρίμ Νταλή, επίσης και εσάς σας καλύτερη η απάντηση ότι δεν καταλαβαίνω πραγματικά γιατί δεν αναφέρεται ποτέ η στατική σημασία του άξονα Λιών Τωρίνου. Δεν καλύπτεται από τα όσα εσείς ε, είπατε, ούτε εσείς από την Ισπανία, ούτε ο κύριος από την Ιταλία. Γιατί είναι το, το, το, το επίκεντρο αυτής της στρατηγικής. Και θα ήθελα λοιπόν να σας ρωτήσω γιατί ποτέ δεν το λέτε. Βέβαια επί 8 χρόνια ασχολούμαι με το θέμα και κάτι ξέρω. Αλλά νομίζω ότι το σωστό θα ήταν να αναδειχθεί αυτός ο στρατηγικός χαρακτήρας από ευρωπαϊκής πλευράς. Η κυρία είστε ευρωβουλευτής. Οπότε σας ρωτώ. Ε, δεν ενδιαφέρεστε για, για αυτή την υπόθεση που αφορά ισπανού Ισπανούς, άλλου ε, Ιταλούς, άλλους Τώρα, για τη χρηματοδότηση. Στις 5 Ιουνίου, δηλαδή πριν από μια εβδομάδα, είχαμε τις δύο χώρες οι οποίες ε, υπέβαλαν την ε, έκθεση πιστοποίησης του κόστους που επιβεβαιώνει τις ε, αξιολογίες που είχαν προηγηθεί. Επιβεβαιώνονται επομένω οι υπολογισμοί που είχαν γίνει για την οριστική εκδοχή του έργου. Επομένως η Επιτροπή με το το 40% Και επίσης αυτή η ειδική επιτροπή που συμπληρωτήθηκε από, από Γαλλία και Ιταλία επιβεβαιώνει το κόστος, τον υπολογισμό του του κόστους και επίσης αναφέρεται σε αυτήν την έκθεση ότι είναι λογικό το αν ξεκινήσει πρώτη εβδόμου του 17 το έργο θα ολοκληρωθεί το 2028-29 με τίποτα σε 30 χρόνια. Και δεν διευθύνεται δυνατότητα ε, εναλλακτικής. Μιλάμε για 3.000 χιλιόμετρα. Βλέπετε τι σημασία έχει το, το έργο. Τώρα τι γίνεται με αυτήν την καταληκτική ημερομηνία. Αυτό φασίστηκαν και κρίθηκαν πάνω από 150 χρόνια. Έχουμε πάνω από 3% κλίση. Θέλει 2-3 ατμομηχανέ τόσο ώστε κανεί να ανέβει κάποια λίγα χιλιόμετρα. Να γιατί δεν λειτουργεί η παραδοσιακή γραμμή. Κάνουμε ό,τι μπορούμε βέβαια στο μεταξύ μέχρι να τελειώσει το έργο. Και εγώ ξέρετε περνάω από εκεί ε, αρκετά συχνά. Οπότε παρακαλώ να είστε λογικοί και εσείς κυρία και εσείς πρόεδρε καταλάβετε ότι αυτή η γραμμή του 1870 δεν είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθεί τη σημερινή ημέρα. Να, το βασικό θέμα. Οπότε όπως είπαμε είναι υποέλεγχο η χρηματοδότηση και οι δύο κυβερνήσεις στο Σαμπερί και στο Τωρίνο έχουν φτιάξει κάποιες εγκαταστάσεις. Έχουμε 150 εργαζομένους στο Σαμπερί και 50 στο Τωρίνο. παρά την αντιπολίτευση στο έργο που όπως τώρα προβάλλετε και εσείς κυρία και εσείς κύριε Πρόεδρε, εσείς, τα έχουν βρει οι κυβερνήσεις. Πρόεδρος. Ευχαριστώ πολύ ενδιαφέρουσα παρουσίαση, πολύ ενδιαφέρουσα προτάσεις. Τρεις παρατηρήσεις για να κλείσουμε. Θα πρέπει εσείς ως πρώην Ευρωβουλευτής να ξέρετε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικές οι γλώσσες εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ο καθένας δικαιούται να μιλήσει τη γλώσσα του. Εάν σας ε, κατακρίνει κανείς επειδή μιλήσατε ε, γαλλικά φερρυπίν ε, στην κυρία Νταλή ή, ολλανδικά στον κύριο που είναι και η μητρική σας γλώσσα, τότε εγώ θα σας περασπιζόμουν γιατί έχετε κάθε δικαίωμα και κοιτάξτε εδώ γύρω είναι και οι διερμηνείς που κάνουν. Βεβαίως για την επόμενη παρουσίασή μου θα το λάβω υπόψη λέει ο κύριος Μπρίνκχορστ. Δεύτερη παρατήρηση. Δεν ήξερα ότι είχαν η Γαλλία και η Ιταλία σχέδιο για τη χρηματοδότηση, για το ότι υπάρχει το σχέδιο της σύραγγας, το ήξερα, αλλά για τη χρηματοδότηση για τα επόμενα 20 χρόνια. Τη στρατηγική ε, σημασία επίσης την αναγνωρίζω, αλλά ε, θα πρέπει να κοιταχθούν οι εναλλακτικέ. Αυτό ήθελα να πω. Σας ευχαριστώ θερμά, θα τα ξαναπούμε φαντάζομαι στην τρέχουσα θητεία. Καλή επιτυχία και καλή διασκέδαση στη δουλειά σας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 Also, meine Damen und Herren, jetzt geht es noch weiter zu unserem letzten Punkt. θέμα, τρίτη αυτή την εβδομάδα. Περιφερειακά αεροδρόμια χρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Με μεγάλη χαρά σας καλωσορίζουμε εδώ. Κύριε Ζωφ Πουφά, Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο και τον κύριο Λουκ Τουζόν, κεφαλή τη ομάδα. Ο κύριο Πουφόν έχει πρώτο το λόγο. Το πολύ δέκα λεπτά. Ευχαριστούμε που ήρθατε και περιμένουμε με πολύ ενδιαφέρον την παρουσίασή σα. Ευχαριστώ και καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Πρόεδρο Κράμερ για την πρόσκληση που μου απέφθηνε τον Ιανουάριο του 2015. Να σας παρουσιάσω την ειδική έκθεση του ελεγκτικού συνεδρίου. Έχει παρουσιαστεί επίσης η έκθεση αυτή το Δεκέμβριο του 2014. Ε, υποδομές λοιπόν αεροδρομίων ε, και ε, απόδοση των επενδύσεων. Αυτός είναι ο τίτλος εκθέσεως. Έχουμε να κάνουμε 2,3 εκατομμύρια άτομα που χρησιμοποιούν περί τα 500 εμπορικά αεροδρόμια της Ευρώπης κάθε μέρα. Οι κύριες ε, πλατφόρμες με το 80% δηλαδή του συνόλου του, της κίνησης σε ευρωπαϊκό επίπεδο ενώ το 4% των επιβατών χρησιμοποιείται περιφερειακά αεροδρόμια. Ο τομέας άμεσα ή έμεσα απασχολεί πάνω από ένα εκατομμύριο εργαζομένους. Τα αεροδρόμια και οι σχετικές εταιρείες συμβάλλουν κατά 140 δις το χρόνο στο ΑΕΠ της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κατά την αξιολόγηση των επιδόσεων των υποδομών, το συνέδριο ασχολήθηκε ιδιαίτερα με την με το εάν έχει αποδειχθεί η ανάγκη για την ανάπτυξη των υποδομών, αν έχουν τηρηθεί τα χρονικά και τα δημοσιονομικά όρια για τις υποδομές και την ε, κατασκευή τους, αλλά και αν αξιοποιούνται αυτές οι υποδομές. Επίσης εξετάζουμε αν η επένδυση μεταφράζεται και σε αύξηση του αριθμού των επεβατών ή και βελτίωση Τη υπηρεσία που προσφέρεται στον επιβάτη. Ουσιώδη ζήτημα για, το, για τον έλεγχό μας ήταν το αν το αεροδρόμιο που χρηματοδοτεί η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι βιώσιμο οικονομικά και αν μπορεί να βοηθήσει να συμβάλλει στη δημιουργία της συνεργασίας. Για να λάβουμε τις σχετικές απαντήσεις λοιπόν σε ερωτήσεις μας, ελέγξαμε 20 αεροδρόμια διαφορετικών κρατών μελών Ισπανίας, Ιταλίας, Ελλάδας, ε, ε, Πολωνίας, Σλοβενίας και είδαμε αεροδρόμια που είχαν λάβει συνολικά 666 εκατομμύρια ευρώ από το Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Ταμείο Συνοχής 400 εκατομμύρια δε ήταν αυτά που ελέγχθησαν δημοσιονομικά ε, και βλέπουμε τις εξής διαπιστώσεις. Πρώτον, υπάρχει ένας λόγος πίσω από τις περιπτώσεις ε, για την ανάπτυξη των υποδομών. Σε 10 από τα 14 αεροδρόμια ε, είχαν υλοποιηθεί έργα κατασκευής τερματικού ενώ στη συνέχεια μόνο 2 από τα 14 χρειάζονταν ε, από ό,τι αποδείχθηκε. Η λειτουργία των δύο αεροδρομίων που χρηματοδότησε η Ευρωπαϊκή Ένωση κατά 11 εκατομμύρια ευρώ δεν χρειάζονταν καν. Επίσης, ε, η επέκταση των διαδρόμων προσγειώσεως και ε, στάθμευσης των αεροπλάνων δεν ήταν αιτιολογημένη σε τρεις περιπτώσεις. Εν όλο το συνέδριο υπολογίζει πως 9 από τα 20 αεροδρόμια που ελέγχθηκαν παρουσίαζαν ε, ένα ή περισσότερα έργα μη χρήσιμα. 629 εκατομμύρια ευρώ δηλαδή, επιδοτήσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης αφιερωμένες στα περιφερειακά αεροδρόμια. Ελέγχθησαν. Δεύτερον, έγιναν τα έργα όπως είχε προβλεφθεί. Ελέγχει το ελεγκτικό συνεδρίο και διαπιστώνει ότι σημαντικές καθυστερήσεις υπήρχαν ως προς την κατασκευή και τελική παράδοση των υποδομών για τα 17 από τα 20 αεροδρόμια που ελέγξαμε. Μέση καθυστέρηση δε ήταν 23 μήνες. Υπέρβαση κόστους είχαμε επίσης σε 9 αεροδρόμια και υπέρβαση κατά 95,5 εκατομμύρια ευρώ των δαπανών από αυτά που είχαν αρχικά προβλεφθεί στον προπολογισμό. Τρίτον, το εύρος της κατασκευής ήταν κατάλληλο. Το ελεγκτικό συνέδριο διαπιστώνει ότι η μέση χρήση των τερματικών ήταν σημαντικά χαμηλότερη από την τιμή αναφοράς για 104 επιβάτες ένα τετραγωνικό μέτρο κατέτος. Μόνο 4 από τα 14 αεροδρόμια έφτασαν στην τιμή αυτή προσέγγιση για το επίπεδο ανάπτυξης που ήταν πραγματικά απαραίτητο δεν είχε καμία σχέση με την πραγματικότητα και μέγα μέρος του προγραμματισμού είχε βασιστεί σε υπερβολικά αισιόδοξε προβλέψεις σχέση με σημαντική αύξηση του αριθμού των επιβατών για το μέλλον. Επίσης αξιολόγησε το Ελληνικό Συνέδριο την, ε, το δυναμικό των διαδρόμων και μόνο 64% των υποδομών που κατασκευάστηκαν αντιστοιχούσε σε πραγματικές ανάγκες. Είχε δημιουργηθεί υπερβολικό δυναμικό δύναμο, δηλαδή σε 11 από τα αεροδρόμια που ελέγξαμε. Εν όλο, 55% από το μισό των κονδυλίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ελέγξαμε, 255 εκατομμύρια ευρώ, είχαν αφιερωθεί σε υποδομές που ήταν άχρηστες και περιττές. Ε, τέσσερα, αξιοποιήθηκαν ε, οι κατασκευές. Μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι το μεγαλύτερο κομμάτι των υποδομών που χτίστηκαν με κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης χρησιμοποιήθηκε. Αλλά 38 εκατομμύρια ευρώ όλο αφιερώθηκε σε δομές και υποδομές που δεν αξιοποιούνταν κατά τη στιγμή του ελέγχου. Πέμπτον, μπορούσαμε να περιμένουμε ότι οι επενδύσεις ε, αντιστοιχούν σε όρους ε, κόστου αποτελέσματος. Ε, Βεβαίω διαπιστώνουμε ότι δεν θα μπορούσαν να υλοποιηθούν παρά μόνο εάν ε, τα αναμενόμενα έσοδα ήταν υψηλότερα στο κόστος. Αλλά συγκρίνουμε το κόστος ανά επιπλέον επιβάτη όταν η ε, επένδυση αποφασίστηκε. Με βάση τελευταίες δηλαδή πληροφορίες που είμαστε θέση μα από τα 10 ε, εκ των 20 αεροδρομίων το κόστο ανά επιβάτη αντιστοιχούσε λίγο πολύ στι προβλέψει για ορισμένα ήταν πολύ ψηλότερο από αυτό που είχε αρχικά προβλεφθεί στο σχέδιο της, του προγραμματισμού, ενώ για 7 ακόμη το κόστος για ε, τον κάθε επιπλέον επιβάτη ξεπερνούσε κατά το διπλάσιο της αρχικής προβλέψης. Έκτον, είναι βιώσιμα τα αεροδρόμια. Για να δώσουμε απάντηση, αναλύσαμε την χρηματοοικονομική κατάσταση των αεροδρομίων. Η ανάλυση έδειξε ότι μόνο 4 από τα 20 ελεγχθέντα αεροδρόμια είχαν οικονομική αποδοτικότητα κατά τη διάρκεια του ελέγχου, κατά την εποχή του ελέγχου. Ε, μπορεί να υπάρξει κάποια εξισορρόπηση οικονομικών όρων ε, μεσοπρόθεσμα, αλλά πολλά από αυτά είχαν σημαντικές απώλειες από το 7 έως το 12. Επίσης δείχνει η έρευνά μας ότι τα αεροδρόμια που είχαν λιγότερους από 100.000 επιβάτες ετησίως σημειώνουν ζημία 130 ευρώ ανά επιβάτη κατά τη διάρκεια της σα περίοδου. Πρόκειται εν γέννη για μικρότερα περιφερειακά αεροδρόμια τα οποία δυσκολεύονται να συνεχίσουν την δραστηριότητά τους ε, χωρίς την κρατική ή τη δημόσια επιχορήγηση. Έβδομον, τι αποτέλεσμα είχαν αυτά τα γεγονότα. Διαπιστώνουμε ότι τα 10 εκ των 20 ελεγχθέντων αεροδρομίων μπόρεσαν να αυξήσουν τον αριθμό των επιβατών τους μεταξυ από το 2007-2013, ότι υπήρξε βελτίωση ως προς την υπηρεσία προς τον επιβάτη, προς τον χρήστη, αλλά περιορισμένη, δεν δημιουργία θέσεων εργασία και οικονομική ανάπτυξη, ε, μπορούν να θεωρηθούν ως ε, αξιόλογοι στόχοι για την επένδυση σε περιφερειακό αεροδρόμιο μένα, αλλά δεν έχει υπολογιστεί το οικονομικό όφελος που προέκυψε. Επίσης υπάρχει έλλειμμα αποδεικτικών στοιχείων που να μας οδηγεί στη διαπίστωση ότι χάρη στην ε, επένδυση σε περιφερειακά αεροδρόμια δημιουργήθηκαν νέες θέσεις εργασίας. Επίσης μπορούμε να πούμε ότι μπορεί να συνδεθούν κάποιες νέες θέσεις εργασίας ε, στο θέμα αυτό, ε, στα αεροδρόμια δηλαδή, να αποδοθούν οι νέες θέσεις εργασίας, αλλά μόνο για τέσσερα αεροδρόμια. Συνολικά λοιπόν, πώς βλέπουμε τα αίτια ε, των ε, διαπιστώσεών μας. Ε, τις έχουμε βέβαια αναλυτικά τα αίτια αυτά, αλλά συνοπτικά μπορώ να σας πω ότι ήταν υπερβολικά αισιόδοξε οι προβλέψει στον οργανισμό των επιβατών. Δεύτερον, ήταν πολλέ οι παρόμοιε επενδύσει σε πολύ κοντινά μεταξύ του αεροδρόμια. Τρίτον, ότι υπήρχε έλλειψη των τονισμού μεταξύ κρατών μελών κατά τη στιγμή όπου οι αποφάσει για την επένδυση ελήφθησαν ένα μόνο από τα πέντε κράτη-μέλη είχε μια μακροπρόθεσμη ε, στρατηγική για την ανάπτυξη των αεροδρομικών υποδομών. Ε, τέταρτον, ε, είχε περιορισμένη γνώση των τεκτενωμένων στο με αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Λειτουργία του συστήματος, λειτουργία του συστήματος για την κατανεμημένη διαχείριση δεν επιτρέπει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ελέγχει και να παρακολουθεί ταυτόχρονα όλε τι επενδύσει των κρατών μελών στον τομέα των αεροδρομίων. Πρέπει να διαπιστώσουμε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν γνωρίζει εν γέννη ποιο λαμβάνει τη χρηματοδότηση και δεν γνωρίζει και για ποιο ποσό. Και έτσι περιορίζεται η ικανότητά της να παρακολουθήσει τις εξελίξεις. Ε, τι συνιστούμε. Συνιστά τα εξή στο ελεγκτικό συνέδριο. Πρώτον, να περιοριστεί η πρικοδότηση από τον Ευρωπαϊκό Προπολογισμό στο μέλλον. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει κατά την προγραμματική περίοδο για το 2014-2020 να ε, στηρίξει μόνο τις υποδομές αλλά και τα κράτη-μέλη αντίστοιχα, τις υποδομές των αδρομίων που έχουν βιωσιμότητα οικονομική και εκεί όπου έχει γίνει η σωστή απόδειξη και ανάλυση των οικονομικών στοιχείων. Αυτό στο στάδιο της έγκρισης και της παρακολούθησης του λειτουργικού σχεδίου από την Επιτροπή και για να αποφευχθεί το υπερβάλλον δυναμικό, το περιττό δυναμικό και η επικάλυψη. Θα πρέπει να γίνουν επιλογές ως προς τις αεροδρομικές ε, αεροπορικές υποδομές και να καταθέσουν εθνικά ή υπερεθνικά περιφερειακά σχέδια ε, αεροπορικών υποδομών τα κράτη-μέλη. Τελευταία παρατήρηση. Σας ευχαριστώ που μου επιτρέψατε να παρουσιάσω την έκθεση αυτή και θα ήθελα τώρα να δώσω το λόγο στον επικεφαλής της ομάδας μας, τον κύριο Λίπτον ο οποίος θα παρουσιάσει ορισμένες παρατηρήσεις για τη μεθοδολογία του ελέγχου μας. Ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα σας. Λέγομαι Λουτιούν και είμαι ο επικεφαλής της ομάδας για τον έλεγχο αυτό. Θα ήθελα στα γρήγορα να σας δείξω μερικές διαφάνειες για να μην έχουμε παρερμηνίες ή παρανοήσεις. Μια και είχαμε την εντύπωση ότι στην προηγούμενη συζήτηση κάτι τέτοιο συνέβη. Ποιο ήταν το, το πεδίο εφαρμογής του ε, ελέγχου μας. Εάν έχετε ερωτήσεις, βεβαίως είμαστε στη διάθεσή σας. Αν σας πω λοιπόν πως ε, καλύψαμε, όπως είπαμε, πέντε κράτη-μέλη, 80% των ε, ποσών που δαπανήθηκαν, 20 αεροδρόμια και για το βήμα ουσιαστικότητα να σας πω πως είχαμε αυτά που βλέπετε στον πίνακα. Αν είχαμε ε, πλήρη ουσιαστικότητα θα είχαμε πει 11 αεροδρόμια στην Ισπανία, οπότε θα είχαμε υπερβολές. Το ε, καλύψαμε με μόλις 8 αεροδρόμια στην Ισπανία. Επόμενο, επιλογή αεροδρομίων. Ποια μεθοδολογία ακολουθήσαμε. Καταρχήν, χωρίσαμε σε τέσσερα επίπεδα όλα τα μεγάλα του Ταμείου Συνοχής. Είναι κομμάτι του πληθυσμού προς έλεγχο, γιατί θέλαμε να αξιολογήσουμε τη διαχείριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Για τα λιμάνια το 2010, τα θαλάσσια, πως δεν ήταν πολύ αξιόπιστη, οπότε τα τοποθετήσαμε στο δείγμα. Δεύτερον, θέλαμε πέντε να γίνουν σε ανάλυση κινδύνου, πέντε τυχαία στο δείγμα και τα υπόλοιπα είναι τα ουσιαστικά αυτά δηλαδή, που εξασφαλιάζουν την ουσιαστικότητα. Για τις πέντε χώρες είχαμε έξι συνοχής και όλα τα υπόλοιπα ακολούθησαν τα υπόλοιπα κριτήρια. Και στα αεροδρόμια μπορώ να σας δώσω λεπτομέρειες αργότερα αν σας ενδιαφέρει. Το ρυθματολόγιο ήταν τριπλό Πρώτο, οι επενδύσεις είναι χρήσιμες, η διαχείριση είναι καλή και απέδωσε το κόστος επένδυση βλέποντας τα παραδοτέα. Κατασκευάστηκαν, χρησιμοποιήθηκαν, είχαν τα αποτελέσματα που ε, προσδοκούσαμε. Ποιος είναι ο αντίκτυπος. Ήθελα να πω δύο λόγια για την κρίση, γιατί και αυτό αντικρούστηκε την τελευταία φορά όταν είπαμε πως είχε περιορισμένες συνέπειες η κρίση. Θα σας δείξω κάποιες διαφάνειες για να σας εξηγήσω. Αλλά η παρουσίαση δεν είναι τέλεια γιατί δεν βλέπουμε εδώ στα δεξιά τι ακριβώς σημαίνουν αυτές οι γραμμές. Μαύρη γραμμή. Δεν φαίνεται εύκολα όλα τα αεροδρόμια στις πέντε χώρες που ελέγξαμε. Μοβ αυξάνεται ε, πολωνικά βλέπουμε εκεί μια συνεχή αύξηση ενώ Εστονία στο Πορτοκαλί ε, κάμψη το 2009 λόγω προβλημάτων με την Air Estonia το βασικό μήνυμα είναι πως εκτός από το 8 και το 9 δεν έχουμε συγκεκριμένες συνέπειες από την κρίση εκτός από την μπλε γραμμή που είναι το 11 που έχουμε τον την τραπεζική κρίση στην Ισπανία. Μετά. Νομίζω πως θα πρέπει να έρθουμε να ελέγξουμε εδώ πέρα την τεχνολογία σας, γιατί δεν ξέρω αν είναι αποδοτική η τεχνολογία που έχετε. Δεύτερον, είναι οι ροές επιβατών στα ελεγχομένα αεροδρόμια, τρεις γραμμές εδώ, η μαύρη, όλα στις 27 χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης, αύξηση 6% μετρήθηκε από το 7 μέχρι το 13, πράσινη γραμμή όλα τα αεροδρόμια στα 5 συγκεκριμένα κράτη-μέλη και η μπλε γραμμή τα 20 υποέλεγχο αεροδρόμια. Τι σημαίνει αυτό? Ίσως στέλνουμε χρηματοδότηση στα λιγότερο αποδοτικά αεροδρόμια. Εκεί καταλήξαμε. Είχαν σχεδιάσει σωστά λοιπόν. Αυτή είναι η απάντηση στην πρώτη ερώτηση. Το βασικό είναι που λέμε για τα 13 από τα 18 είχαμε σημαντικές επικαλύψεις στους ε, επιβάτες που προσπάθησαν να προσελκύσουν. Είχαμε και δύο νησιωτικά, η Λαπάλμα και η Φόρτα Βεντούρα, που αποτελούν ένα παράδειγμα και θα σας δείξουμε τι συνέβη. Χρησιμοποιούμε στοιχεία της Eurostat όπου μας δίνουν τα στατιστικά δεδομένα τα πιο πρόσφατα και μια χαρτογράφηση των αποστάσεων για να μπορούμε να καταλήξουμε. Για τη διαχείριση λίγα έχω να πω, δηλαδή το πιο σημαντικό είναι το πρώτο εκεί στη γραμμή. Η χρηματοδότηση έχει ως σκοπό να δαπανηθούν κονδύλια, όχι να έχουμε απόδοση και αποτελεσματικότητα. Σε δύο κράτη-μέλη τουλάχιστον η χρηματοδότηση ήταν πιο σημαντική για το κράτος από τα ενδεχόμενα αποτελέσματα. Τρίτον, και εδώ είχαμε αρκετές πληροφορίες, είχαμε αρκετές περιπτώσεις με καθυστερήσεις, αύξηση και υπέρβαση κόστους, οικοδομήσεις κτηρίων που δεν χρειάζονται, περιορισμένη βελτίωση της ποιότητας. Δύο συγκεκριμένες διαφάνειες θα σας δώσουν μια εντύπωση για το πώς μετρήσαμε τις ανάγκες μας. Αυτή είναι μια θετική εικόνα γιατί πριν δούμε αν έχουν εκτιστεί τερματικοί σταθμοί, είπαμε δείξεις αναφοράς 104 επιβάτες ανά τετραγωνικά μέτρο ο, χωρητικότητας και αυτό σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη αναφοράς της ΙΑΤΑ. Άρα λοιπόν η κατάνοια είναι μια προφανής περίπτωση όπου ο κόσμος έκανε ουρά εκτός τέρμιναλ και χρειάστηκε να στήσουν ένα λιόμενο για να καλύψουν τις ανάγκες για τον Πανταχώς δεν χρειαζότανε. Αλλά αν δούμε τι οικοδομήθηκε και πολλές φορές είναι τόσο υπερβολικό το μέγεθος που δεν καταφέρνουν ούτε να πετύχουν το 50% του δίκτυου αναφοράς. Νομίζω ότι αυτό είναι και ο πιο εύκολος τρόπος να το δει κανείς. Περιορισμένα λοιπόν ποιοτικά αποτελέσματα, φτωχή βιωσιμότητα, πολύ περιορισμένη επίπτωση που να τακμηριώνεται. Οπότε υπάρχει πρόβλημα. Λοιπόν, so we μηνύματα κλειδιά. Οι δύο συστάσεις που έχουν ήδη ε, παρουσιαστεί από τον κύριο Πουφών είναι οι εξής. Ευρήματα παρόμοια με αυτά του ελέγχου θα μπορούσαν να έχουν διαποσχεθεί και σε άλλα κράτη-μέλη υπό έλεγχο. Κύριε Πρόεδρε, εσείς αναφερθήκατε στη χώρα σας, αλλά υπάρχουν και άλλοι. Στη μελέτη μας μάθαμε πως η επικάλυψη, η η περιορισμένη χρήση είναι προβλήματα και σε άλλα κράτη-μέλη. Το μήνυμα αυτό θα πρέπει λοιπόν να το κατανοήσουν όλοι. Δεύτερον, αυτό που λάβαμε υπόψη είναι όχι μόνο τις δημοσιονομικές συνέπειες, αλλά και τα οικονομικά αποτελέσματα, αλλά και την προσβασιμότητα. Αυτό που προσπαθούμε να αποφύγουμε όσο μπορούμε στη μεθοδολογία μας είναι τα νησιά. Γιατί δεν μπορεί να κολυμπήσει κανείς ένα νησί ή έχει αεροδρόμιο και λιμάνι ή τίποτα. Οπότε όπου μπορούσαμε τα βγάλαμε από τον πληθυσμό. Τα μόνα που ήταν υποχρεωτικά να ε, εξεταστούν ήταν η Βεντούρα και Λας Πάλμας, γιατί εκεί βέβαια ήταν πολύ μεγάλα τα έργα αυτά. Τέλος, έχουμε ένα μακρύ κατάλογο του τι θα πρέπει να κάνουμε έτσι ώστε να είναι λογικά τα κονδύλια που δαπανώνται. Λοιπόν, προτεραιότητες, μακρόπνο σχεδιασμός, αξιολόγηση κόστους, σχέση κόστους οφέλους, η οποία καμιά φορά δεν λαμβάνει υπόψη τα πραγματικά κόστη, εξελίξεις σε ανταγωνιστικά συγκοινωνικά μέσα, υψηλής ταχύτητας τρένα για παράδειγμα, και διασύνδεση με λιμένες, για να δούμε τι έχει επενδυθεί εκεί. Και αν είναι όλα πράσινα τα κουτάκια, τότε θα πρέπει να επενδύσουμε και όχι να σταματήσουμε τις επενδύσεις αυτές. Εάν έχετε ερωτήσεις, με χαρά να απαντήσω. Ευχαριστώ και εγώ και τους δύο μελητές. Πολύ σοβαρή έρευνά σας θα μας ε, δώσει, μας δίνει πολλά στοιχεία. Η κυρία Κλού έχει το λόγο παρακαλώ. Ε, Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε τους ε, δύο κυρίους για τις εισηγήσεις τους. Έχετε δίκιο πρόεδρε, πολλά μπορούμε να μάθουμε και είναι ενδιαφέρον να ακούμε την μεθοδολογία που χρησιμοποιείται για τα αεροδρόμια. Βλέπουμε αυτή την έκθεση, πρόκειται για 28 κράτη-μέλη. Δεν συμμετέχουν μόνο 5. Γι' αυτό είπατε ότι 78%, 80% χρησιμοδότηση αφορά αυτές τις χώρες. Είναι σημαντικό. Να δούμε επομένως πώς δαπανήθηκαν ε, τα χρήματα, πώς μπορούσαν να δαπανηθούν καλύτερα, τι καθυστέρησες έχουμε. Πολύ σημαντικό αυτό που θα πρέπει ο πλευρά οικονομικού ελέγχου να το προσέξουμε. Πολλά ε, σήμερα δεν μπορούμε να εξαγαγούμε. Χρειάζεται ένα αεροδρόμιο. Τι υπάρχει το αεροδρόμιο, τι διευκολύνσεις υπάρχουν. Έχουμε στοιχεία δημιουργούν θέσεις ε, απασχόλησης. Έχουμε νομίζω κάποια, κάποια στοιχεία, πόσο συνέβαλαν τα αεροδρόμια. Έχω εδώ κάποια στοιχεία. 124 θέσεις για κάθε 100.000 επιμετρήθηκα. Και σε σχέση με το ΑΕΠ. 10.000 επιβάτες άκουσαν το ΑΕΠ κατά 0,5%. Να επομένως κάποια στατιστικά στοιχεία που μας δώσανε. Υπάρχει συμβολή βοηθάτε το ΑΕΠ και η απασχόληση. Είναι επομένως πολύτιμα αυτά τα αεροδρόμια που συζητούμε. Καλό το να έχουμε τα στοιχεία και τα δεδομένα, αλλά είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει ε, σύνδεση μεταξύ των αεροδρομίων ε, η σύνδεση της περι... κάποιες περιφέρειες με το αεροδρόμιο. Μιλάμε για κόμβους. Αυτό είναι σημαντικό για τον τουρισμό και όχι μόνο. Ε, βέβαια, εάν κανείς δεν έχει αεροδρόμιο, δεν θα έχει επενδύσεις, δεν θα έχει τουρισμό. Επομένως, θα πρέπει να δούμε τα πραγματικά στοιχεία. Τα γεγονότα, πώς θα μπορέσουμε να δημιουργήσουμε το, το αναγκαίο κοινωνικο-οικονομικό πλαίσιο. Μέσα εκεί θα πρέπει να κινηθούμε και να το σκεφτούμε. Βέβαια, λαμβάνω υπόψη ότι έχουμε κάποια, α, κάποια οικοδομήματα, κάποια κτίρια που υπερβαίνουν τον προϋπολογισμό. Από την δική μου εμπειρία, από όσα ακούω, για την περίοδο 14-20, Υπάρχει πίεση από την ε, ε, Επιτροπή. Πώς δαπανήθηκαν οι πόροι. Τι γίνεται με αυτά τα αεροδρόμια. Πρόκειται για δημόσιο χρήμα. Αν επομένω χρειάζονται τα αεροδρόμια, αν έχουμε επικάλυψη, αν δημιουργούν θέσει απασχόληση και έχουμε αυτέ τι κατευθυντήριε γραμμέ. Τι γίνεται σε σχέση με τα άλλα μέσα μεταφορά, ε, οδικά, σιδηροδρομικά Υπάρχουν ένα σωρό παράμετροι. Φορτεβεντούρα, Πάλμα. Αν δεν είχαν αεροδρόμιο θα υπήρχε καμία δραστηριότητα. Φυσικά και χρειάζονται και διασυνδέσει μεταξύ διαφορετικών ειδών μεταφοράς. Και ακόμη πιο σημαντικό είναι βέβαια να υπάρχει εποπτεία, έλεγχος των δαπανωμένων κονδυλίων. Να μην υπάρχει κακή χρήση αυτών. Μην υπάρχουν επίσης επικαλύψεις. Πάντως είναι πάρα πολύ σημαντικά τα περιφερειακά αεροδρόμια για την ε, Ήπερο, Ήπεθρο, συγγνώμη, για τις αγροτικές περιοχές. Και σας τα λέω αυτά μια που είμαι Ιρλανδέζα. Πολύ σημαντικό. Δεν θα είχαμε ε, διασύνδεση χωρίς αεροδρόμια. Danke sehr. Jetzt Ines κυρία Ευχαριστώ, πρόεδρε. Τι είναι αυτό, κάτι σαν ομπρέλα, σαν κάλυψη που προσπαθεί να κάνει τώρα ε, το ελεκτικό συνέδριο για να υπεραμεινθεί αυτού του οικονομικού ελέγχου που ε, βάσει ε, της ε, ε, δειγματοληψίας μας δείχνει το θέμα είναι ότι θα μπορούσαμε να έχουμε καλύτερο οικονομικό έλεγχο και να έχουμε πιο ευρεία δειγματοληψία. Έτσι γίνεται στο Νότο με τους πόρους συνοχής. Οπότε έχουμε και κάποια αεροδρόμια που έχω την τύχη και βέβαια είναι πιο ευθύς αυτά ο κύριος Κράμερ από άλλους. Ξέρουμε ότι υπάρχουν προβλήματα σε ένα αεροδρόμιο και τα, τα τελικά τα πιο μεγάλα προβλήματα βρίσκονται στο αεροδρόμιο της πρωτεύουσας του κόσμου, δηλαδή του Βερολίνου. Επομένως, ήταν πάρα πολύ το πω διπλωματικά περίεργη δειγματοληψία του ελληνικού συνεδρίου. Θα πρέπει κάποια στιγμή να κάνει οικονομικό έργο αυθεντικό. Δεν είναι μόνο να ασχολούμαστε με τον ε, Νότο και δηλαδή σε δύο νησιά που έχουν εξυπηρέτηση υποχρεωτική Πάλμα και Φορτεμιδούρα. Είναι υποχρεωτική η δημόσια κάλυψη εκεί. Μιλάμε όμως επίσης και για τουριστικά κέντρα. Εκεί που υπάρχουν ε, τουρίστες από παντού. Και βλέπουμε εδώ κάποιες φωτογραφίες που είναι συγκλονιστικές. Τώρα, όσον αφορά την κρίση. Ξεκινάμε το 2007. Τότε ξεπίδησαν όλα. Μετά ξέσπασε η κρίση την επόμενη χρονιά. Και λέμε για τον Νότο, για την Μεσόγειο. Είχαμε τα γεγονότα στην Τίνιδα. Οπότε ωφεληθήκαμε εμείς τουριστικά. Βέβαια δεν είναι σωστό αυτό να φαίνεται στην τραγωδία του άλλου. Πάντω έχουμε κάποια αεροδρόμια που χάσανε μέχρι και 20 εκατομμύρια. Αυτό δεν εμφανίζεται εδώ. Έχουμε κάτι άλλα αριθμητικά στοιχεία. Αλλά θα ήθελα να ξέρω πόσο χάσανε σε αυτή την περίοδο από το, από το 7 μέχρι την περίοδο, την ημερομηνία που τέλειωσε ε, ο έλεγχος, γιατί τα, τα σκόντασε τα αεροδρόμια η κρίση. Τι έγινε με την ανάπτυξη και τον τουρισμό. Εσείς λοιπόν μένετε σε αυτά τα στοιχεία και λέτε ότι δεν έχει σχέση με την κρίση, μα φυσικά και είχε. Επομένως, τα στοιχεία αυτά είναι τρομερά. Χάσαμε 20, 20 εκατομμύρια ε, συνολικά επιβατών. Επομένως, 11 εκατομμύρια χάσαμε ε, μόνο στην Μαδρίτη. Επομένως, τι λέμε, θα πρέπει να μειωθεί η χρηματοδότηση κάποιων αεροδρομίων. Δεν λάβετε υπόψη το ψήφισμα Μπράντμπορν του 2012 εδώ στην Επιτροπή αυτή για τα περιφερειακά αεροδρόμια. Αυτό, όσον αφορά την μέτρηση των αποτελεσμάτων, είναι σημαντικό. Όχι μόνο το κέρδος αν επιβάτη μέσα στην κρίση και μιλάμε για ε, έντονο εποχιακό χαρακτήρα που έχουν ε, τα έσοδα σε κάποια αεροδρόμια. Επομένως, γιατί αγνοήσα την έκθεση για αυτά τα αεροδρόμια σε πολλά μέρη, αλλά ε, σε πολλά μέρη έχουμε τον τουρισμό και πώς θα επιζήσουν αυτά τα ε, μέρη που έχουν πλήγει από την Τρόικα. Λέτε ότι υπάρχει διασπάθηση πόρων, αλλά σε κάποια μέρη λόγω της γεωγραφικής διαμόρφωσης μόνο με αεροδρόμιο μπορούν να έρθουν και να φύγουν οι τουρίστες. Μα να διαλέγετε την Πάλμα και την Φορτιβεντούρα για παράδειγμα είναι τρομερό. Ο πρόεδρος. Κύριος Νίλσον. Ευχαριστώ πρόεδρε. Ναι. Θέλω να αφαιρθώ σε κάτι που έλεγε ένας δήμαρχος πριν από χρόνια, ότι δεν πρέπει πάντα να επικοινωνούνται τα πάντα. Αλλά αυτό που θέλουμε να πούμε εδώ είναι ότι θα ήταν καλό να ξέρουμε η Επιτροπή τι έχει να σχολιάσει για όλη αυτή την υπόθεση. Και πάντα με το βλέμμα προς τα μπρος. Τα περιφερειακά αεροδρομία είναι άκρο σημαντικά. Το δέχομαι και εγώ το υποστηρίζω. στην Επιτροπή των Περιφερειών Σύστημα για Περιφερειακή Πολιτική και εκεί ήμουν και εγώ μέλος. Είναι ένα σαφές παράδειγμα τα περιφερειακά αεροδρόμια για την υλοποίηση της πολιτικής της συνοχής. Και πολύ συγκεκριμένα υλοποιούνται αυτά στα περιφερειακά αεροδρόμια, όχι μόνο από στρατηγικής 2020, αλλά γενικά για την ανάπτυξη μιας περιφέρειας. Πρόκειται για στρατηγικά σημαντικές ε, επενδύσεις που χρειαζόμαστε για να προωθήσουμε την ανάπτυξη. Μπορεί να μην ζουν τόσο πολλοί κάτοικοι σε μια περιφέρεια. Μπορεί να μην είναι δυνατόν να καταστεί βιώσιμο χωρί υποστήριξη το αεροδρόμιο, ακριβώ γιατί είναι περιορισμένο ο αριθμό των κατοίκων που θα το χρησιμοποιήσουν. Άρα χρειάζεται ε, υποστήριξη και από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από τι κυβερνήσει. Δεν πρέπει να λησμονούμε ότι αυτοί οι οποίοι δραστηριοποιούνται σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο βλέπουν το σημαντικό ρόλο των περιφερειακών αεροδρομίων. Αλλά περιμένω να ακούσω τις απαντήσεις της Επιτροπής. Έχει γίνει συζήτηση για τις κρατικές επιδοτήσεις. Η οποία κατέληγε πάντα στο ότι δεν επιτρέπονται οι κρατικές ενισχύσεις. Αν και όταν γίνονται επενδύσεις σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο είναι πολύ καλύτερες οι δυνατότητες πρόσβασης. Γι' αυτό έχουν μεγάλη σημασία αυτά τα περιφερειακά αεροδρόμια. Ο Πρόεδρος, ευχαριστώ θερμά και ρητά για την έκθεση. Πρέπει να μάθουμε, να μαθαίνουμε και από τα σφάλματα. Λέμε για κρίση και κρίσεις. Λέμε ότι πρέπει να ε, διευρύνεται το δυναμικό στα περιφερειακά αεροδρόμια, όπου χρειάζεται όμως. Για παραδείγμα, το αεροδρόμιο Βερολίνο-Τέγκελ ε, οικοδομήθηκε το 2000 και τώρα έχει 70 εκατομμύρια ε, επιβάτες. Ε, άρα υπάρχει το δυναμικό και δυνατότητα της ανάπτυξής τους. Δεν μπορούμε επίσης να πούμε ότι δεν θα κατασκευάσουμε αεροδρόμια για περιφερειές απομακρυσμένες ή νησιωτικές, γιατί εκεί χρειάζεται η διασύνδεση, χρειάζεται να εξασφαλιστεί σε αυτό, δεν θα φέρω αντίρρηση σε επιδοτήσεις. Πρέπει όμως να κοιτάξουμε ποιες είναι οι περιτές επενδύσεις, οι οποίες έγιναν μόνο και μόνο γιατί κάποιος τις οραματίστηκε. Και είναι τεράστια αυτά τα οράματα στις ε, ενέργειες μεταφορές. Ενέργειες μεταφορές που χρηματοδοτούνται με 30 δις από τον Ευρωπαίο Φορολογούμενο κατέτος, γιατί οι εταιρείες δεν πληρώνουν κυροζήνη, φόρο κυροζήνης, δεν πληρώνουν ε, φόρο προσθέμενης αξίας, ενώ όλοι οι άλλοι οφείλουν να, πληρώνουν. 30 δις ευρώ το χρόνο, χάρη σοφίες, ε, χάρη στα οποία και παρά τα οποία παραμένουν να έχουν ελλείμματα ορισμένες εταιρείε. Το Castle Carlton, παραδείγματι, αεροδρόμιο με 29 εκατομμύρια κόστο στη Γερμανία, με 1,5 ε, ώρα απόσταση από το αεροδρόμιο της Φραγκφούρτης, ε, το Castle, σιδηροδρομικός, κατασκευάζεται με 370 εκατομμύρια κόστος ένα αεροδρόμιο στο Κάσλ. Ε, μετά, μεταξύ Ζάρμπρουκεν και Τσβάιμπρουκεν, 30 χιλιόμετρα αεροδρόμια τα οποία είναι ελληματικά, αλλά μια και δεν υπάρχει έννοια εθνικών αεροδρομίων στη Γερμανία, και αφού το Σαρμπρούκεν ανήκει στο, στο Σάρλαντ και στην Ρινανία Παλατινάτο το άλλο αεροδρόμιο, το κάθε κρατήδιο αφού είναι ομοσπονδιακές οι δομές στη Γερμανία φτιάχνει και επιδοτεί το δικό του αεροδρόμιο ενώ θα μπορούσαμε μέσα σε μια-δύο ώρες να είχαμε φτάσει ε, με το τρένο, με ένα τεζεβέ παραδείγματι μέχρι το Παρίσι ή οποιοδήποτε άλλο μεγάλο διεθνέ αεροδρόμιο. Λοιπόν, εκεί πρέπει να γίνεται η επιλογή των ε, ενισχύσεων και των σχεδίων. Το 90% των μεγάλων σχεδίων στις ε, μεταφορές δεν έχουν καμία ε, θεώρηση μεταφορών, απλώς προκύπτει ως υποστήριξη των λόμπι των μεταφορών, για να μην πω και των τραπεζικών λόμπι. Και το λέω διότι υπάρχει ανάλυση του Πανεπιστήμιου της Δρέσδης. Ξέρετε, εκεί υπάρχει ένας δακτύλιος αυτοκινητοδρόμου περιφερειακού γύρω από μία πόλη χωρίς να έχει σημείο εισόδου και εξόδου. Το, το τούνελ Ζέγγελρινγκ στην Αυστρία. Εάν κατασκευαστεί και το ξαναμπαζώσουν μετά, πάλι θα έχει θετικό απολογισμό. Είναι σαν να σας λέω εγώ ότι χτίζω αυτό εδώ το κτίριο, το, κατα... το, το γκρεμίζω μετά και βγάζω πάλι θετικό απολογισμό. Αυτή είναι η ανάλυση που γίνεται. Όχι λοιπόν, πρέπει να κοιτάμε όταν γίνεται ε, η κατασκευή ενός έργου τι είδους συνέπειες θα έχει για το μέλλον. Και αυτές να είναι ο θετικός απολογισμός. Με βάση αυτές να έχουμε το θετικό απολογισμό. Όχι να λέμε κατασκεύασα θέσεις εργασίας και μετά τον γκρεμίζω το έργο. Πιο χρήσιμους τρόπους θα είχαμε να δώσουμε τα χρήματά μας. Για τις επιδοτήσεις, ναι, για τις απομακρυσμένε περιοχές. Σουηδία, Φιλανδία, νησιά, ναι, ορισμένα νησιά, να τις υποστηρίξουμε και να τις πούμε και επιδοτήσεις. Αλλά μεταξύ Βερολίνου και Μπρέσλαου δεν, δεν προχωράει η κατασκευή των σιδηροδρόμων γιατί δεν επιτρέπονται και δεν γίνονται, δεν δίνονται επιδοτήσεις. Ενώ οποιοδήποτε μικρό αεροδρόμιο, εάν σταματούσε, θα μπορούσε να χρηματοδοτήσει αυτή τη σιδηροδρομική γραμμή. Άκουσα ότι μόνο 4 από τα 20 περιφερειακά αεροδρόμια έχουν αποδοτικότητα. Να σας πω ποια είναι η κατάσταση στη Γερμανία. Και δεν μιλάω μόνο για το νέο αυτό αεροδρόμιο του Βερολίνου, του Σόνεφελτ. Έχουμε 23 διεθνή αεροδρόμια στη Γερμανία, εκ των οποίων τα 17 είναι ελληματικά. Έξι μόνο φέρνουν κέρδος ή, εν πάση περιπτώσει, ίσως το κόστος τους. Με, με αυτά τα στοιχεία είναι δυνατόν να λέμε χρηματοδοτούμε ό,τι να είναι δεν πρέπει να κοιτάξουμε πόσα, πόσα έλλειψη έχουμε για το σιδηροδρόμο στην Ισπανία, α πούμε, ή στην Σουηδία. Χρήματα που θα μπορούσαν να πάνε σε άλλου τρόπου μεταφορών σε όλα τα κράτη. Και αυτό δεν είναι θέμα μόνο των νότιων αεροδρομίων. Δεν ήξερα άλλωστε ότι και η Εστονία ανήκει στην Νότια Ευρώπη. Και καινούριο μου φαίνεται αυτό αλλά και αυτή έχει προβλήματα. Α σταματήσει λοιπόν αυτή η κατάσταση, γιατί δεν είμαι διατεθειμένο εγώ να δίνω τα χρήματα του Ευρωπαίου Φορολογούμενου, παρά μόνο είναι για έργο αποδοτικό. Όχι γιατί κάποιο κάποια μέρα ορειρεύτηκε και οραματίστηκε κάτι και μόνο για το όρομα όραμα κάποιανού θα δίνουμε τα λεφτά. Πρέπει να γίνεται πιο σοβαρά η δουλειά και γι' αυτό ερωτώ πώ συνεχίζουμε, τι κάνουμε από εδώ και πέρα. Πολλά κράτη-μέλη πολύ ευχαριστώ θα πάρουν τα ευρωπαϊκά κονδύλια για να στηρίξουν την ε, εγχώρια κατασκευαστική βιομηχανία. Αλλά όταν έχουμε τέτοιου είδους προγνώσεις, οι οποίες επιτοπλίστων ε, ξεχνάνε σχέση κόστους αποτελέσματος, δηλαδή κοιτάνε μόνο το τι θέλει η πολιτική, που εκφράζεται τότε ως φθηνό έργο, ε, και τι δεν θέλει που μετατρέπεται σε ακριβό έργο. Η Στουτχάρδη τίποτα, τζάμπα σχεδόν μας το παρουσιάσανε για να χρηματοδοτήσουν με 10 δισεκατομμύρια τον υπόγειο εκείνο σταθμό <coughs> ε, το σιδηροδρομικό σταθμό της Στουτχάρτης. Γιατί το θέλανε. Ε, πρέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να έχει τη δυνατότητα να ανακτήσει τα κονδύλια, να τα απαιτήσει και πάνω απ' όλα να γίνεται από την αρχή σωστά ο υπολογισμό. Αυτή είναι η ευθύνη μα. Και τι έχετε να πείτε εσεί σαν συνταγή μετά την ανάλυση για το μέλλον, τι πρέπει να κάνουμε για να αποφύγουμε τέτοια φαινόμενα. Μπορείτε να μας απαντήσετε μέσα σε 12 λεπτά. Ευχαριστώ πολύ. Που... Ε, ε, να σας πω το εξή. Ε, για τις ερωτήσεις που μας έκανε η κυρία Κλού να δώσω κάποιες πρώτες απαντήσεις. Είχαμε καθυστερήσεις. Είχαμε καθυστερήσεις στην κατασκευή και στην παράδοση σε 27 από τα 21 αεροδρόμια. Και 14 αεροδρόμια ξεπέρασαν τα χρονοδιαγράμματα τα οποία είχαν προβληθεί κατά ένα χρόνο. Δηλαδή είχαμε καθυστερήσει μέχρι 23 μήνες. Και κύριε Πρόεδρε, ναι, συμφωνώ μαζί σας, χρειαζόμαστε θέσεις απασχόλησης και ξέρω ε, γιατί τα είπατε αυτά και εσείς και οι συναδελφοί σας. Όμως, τι γίνεται μετά. Ωραία. Το ζήτημα δεν είναι μόνο να δημιουργήσουμε θέσεις εργασίας, αλλά και να τις διατηρήσουμε μέσω των κερδών των αεροδρομίων. Έτσι θα γίνει. Μέσω των ε, αερομεταφορών. Το ιδανικό θα ήταν αυτό, όχι μέσω άλλες ε, χρηματοδότησης. Ως γνωρίζω τι σημαίνει περιφερειακό αεροδρόμιο. Εγώ χρησιμοποιώ το Σαρερουά και τη Ράινερδο και πολύ καιρό και είμαι πολύ ικανοποιημένος από την ε, υπηρεσία που μου προσφέρουν. Ακούσαμε και κάποια σχόλια από την κυρία Γιάλα Σέντερ. Τι να πω. Όταν κοιτάξαμε το δείγμα και επιλέξαμε τα αεροδρόμια, έξι από τα αεροδρόμια εκπροσωπούν τα μεγάλα έργα που χρηματοδοτήθηκαν από το Ταμείο Συνοχής. Και τα υπόλοιπα τα επιλέξαμε, μάλλον πέντε ήταν ε, αξιολόγηση κινδύνου και πέντε ε, ε δείγμα, ε, δείγμα. Και πέντε ήταν αυτά τα οποία ε, ήταν τα πιο δαπανηρά. Δίκιο έχετε, δεν μπορεί να επισκεφθεί κανεί ένα νησί αν δεν έχει αεροδρόμιο. Πάντως έγινε μια συζήτηση στην Επιτροπή Κοντ και εκεί τι μας είπατε κυρία Γιάλα Σέντερ, μας είπατε τι συμβαίνει με το αεροδρόμιο στη Μούρσια. Εκεί έχουμε μια πολύ περίεργη κατάσταση όπου χρειάζεται οι επιβάτες που ταξιδεύουν να περάσουν από εκεί γιατί ας πούμε κάνουν μεταμόσχευση καρδιάς. Ξέρουμε τι συνέβη το 2007. Ξέρουμε τις συνέπειες που είχε η κρίση στην κατασκευή αεροδρομίων. Το 2007 εγώ πήγα στη Μαδρίτη. Μιλήσαμε εκεί στους αντιπροέδρους και ευχαρίστησαν τους Ρουμάνους εργάτες, τους οικοδόμους, γιατί συνεισέφεραν στην οικοδομή στην Ισπανία με αύξηση του ΑΕΠ αλλά θα το αφήσω εδώ και θα δώσω το λόγο στο συνάδελφο μήπως και αυτό συμπληρώσει. Στα γρήγορα να πω πως εντάξει, οι θέσεις εργασίας είναι σημαντικές, αλλά στον έλεγχό μας είδαμε πως πολύ λίγες ε, δόθηκαν. Οπότε δεν νομίζω ότι ήταν αυτό ο λόγος για τον οποίο χτίστηκαν τα αεροδρόμια. Για μεγαλύτερο δείγμα μπορούμε. Αλλά και τότε θα ήταν παρόμοια τα ευρήματα που είχαμε αυτά που έχουμε σήμερα. Για, το, για τη Φόρτα Βεντούρα και τη Λαπάλμα, ναι, εντάξει, υπάρχουν τουριστικά αξιοθέατα και δεν είμαστε κατά αυτών των επενδύσεων, όμως έχουμε τόσα τόσο υπερβολικές επενδύσεις σε χώρους και εγκαταστάσεις που σε κάποιο τμήμα σε, και για να κρατήσουν χαμηλό το κόστος συντήρησης κλείνουν και χώρους από το αεροδρόμιο πολλές φορές Οπότε νομίζω ότι αυτό δεν είναι η βέλτιστη χρήση των ε, πόρων των φορολογουμένων. Ποιο είναι το κόστος που επιβαρύνει το φορολογούμενο. 7 από τα 20 δεν θα φτάσουν καν στο σημείο του ισοσκελισμού, της αποπλήρωσης, δηλαδή της επένδυσης. Αυτή είναι μια πολιτική απόφαση που λαμβάνεται σε κάθε περίπτωση και ναι, είναι καθολικό το θέμα, είναι μια συζήτηση όταν ξεκινήσαμε τον έλεγχο στο Λουξεμβούργο. Είχαμε τη Φραγκφούρτη, Φραγκφουρτ Χάν, Λιέγη, Σαρλερουά, Λουξεμβούργο, Πίτμπουργκ, κοντά στο Μέτς, τοπικά αεροδρόμια που κατασκευάστηκαν και έχουν τα ίδια προβλήματα. Ίσως λοιπόν χρειάζεται να γίνει κάποια, κάποιος εξορθολογισμός και από τις πέντε χώρες οι τέσσερις δεν είχαν μακροπρόθεσμη στρατηγική σχεδιασμού αεροδρομίων και μία χώρα είχε τέλος πάντων κάποιο είδος στρατηγική παρόλο που δεν ήταν περίφημη. Θα πρέπει λοιπόν το μήνυμα αυτό να το ακούσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και να ξεκινήσει με την εκ των προτέρων ερεσιμότητα έτσι ώστε να εξορθολογήσει στην επόμενη περίοδο τα θέματα αυτά. Ευχαριστώ. Σάμον Μπρέν, Κομισιόν. Αν έχετε κάτι να πείτε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σαν πριν ονομάζομαι και είμαι ο επικεφαλή του Τμήματο για τα αεροδρόμια όσον αφορά τη Γενική Διεύθυνση για Μεταφορέ και Κινητικότητα. Θα είμαι σύντομο για να απαντήσω σε κάποια από αυτά τα οποία αναφέρθηκαν ε, ότι απαντούμε ε, σε, σε έγγραφο που προσαρτάται στην έκθεση. Δεν συμβαίνει πάντα αυτό, δηλαδή να έχουμε πρόβλημα στη χρήση των πόρων για την υποδομή. Είπαμε ότι έχουμε κάποιες αλλαγές ε, για την περίοδο 14 έως 2020. Είπαμε ότι θα πρέπει να εστιάσουμε προσοχή μας σε ασφάλεια και περιβάλλον. Επίσης ε, προσέχουμε το τι γίνεται με τα κράτη-μέλη όσον αφορά τα αεροδρόμια που ανήκουν στο διευρωπαϊκό δίκτυο. Ε, αυτό το οποίο χρειάζεται είναι να υπάρχει αυτή και των προτέρων αιρεσιμότητα για την χρηματοδότηση και επίσης όσον αφορά τα βασικά πρόγραμματα και έργα και σχέδια η αναφιόρηση ποιότητας είναι κάτι το οποίο ε, πρόκειται να καθιερωθεί και αυτές είναι οι βασικές μεταβολές για την επόμενη περίοδο ούτως ώστε να μπορέσουμε να ε, επιλύσουμε αυτά τα προβλήματα τα οποία δικαιολογημένα επισημαίνει το Ελληνικό Συνέδριο. Τώρα έχω άλλα δύο ζητήματα τα οποία θα πρέπει να τα θίξουν. Πρώτα το θέμα του κατά πόσο υπάρχει κέρδο, αν είναι επικερδίτερα αεροδρόμια. κάποια άλλα στοιχεία έχουμε αυτό το 44% ε, ότι είναι επιζήμια αεροδρόμια. 75% αυτά που έχουν λιγότερο από ένα εκατομμύριο επιβάτε ε, είναι ζημιογόνα. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι όλα αυτά υποστηρίζονται από τον κρατικό κορδόνα, αλλά υπάρχουν κάποιες περιπτώσει δύσκολες, κάποια μικρότερα αεροδρόμια και υπάρχουν κάποιες ε, άλλες πολιτικές, όπως η πολιτική της Ένωσης για τις κρατικές ε, ενισχύσεις. Ε, έχουμε το πρόγραμμα Κέσσερ που βοηθά τα, τα μικρότερα αεροδρόμια. Πάρα πολύ σημαντικό να υπάρχει αυτή η βοήθεια και είπε και κάτι η κυρία Σέντερ που το τονίσατε στην εκθεσή σας για το περιφερειακό εδώ στο Κοινοβούλιο. Τώρα επίσης τελευταία, η φύση των επενδύσεων είναι εξορισμού κάτι το μακρόπνο. Είναι δύσκολο επομένως να κάτσουμε αυτό να το κατα... κατατάξουμε στον χρόνο. Πρόκειται για κάτι το οποίο εξελίσσεται ανάλογα με την εξέλιξη της κυκλοφορίας του αεροδρομίου. Ο Πρόεδρος. Ευχαριστώ και για την τοποθέτηση. Για όλες τις παρουσιάσεις και τη συζήτηση ήταν συναρπαστική, όπως πάντα. Σας ευχαριστώ για την φορά που ήρθατε και κυρίσω το πέρα συνεδρίασης για σήμερα. Και πάμε για την προετοιμασία του αυριανού τριμερού διαλόγου.